Καλησπέρα, ας ξεκινήσουμε την απογευματινή συνεδρίαση. Χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη συνεδρίαση που έχουμε περί ανθρωπιστικής βοηθείας και το μέλλον αυτής της ανθρωπιστικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε τον Επίτροπο τον κ. Στυλιανίδη μαζί μας. Χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Έχουμε δικαιωμένου ομιλητές. Θα δώσω το λόγο στον Ερίκε Γκερέρο Σαλόμ, ο οποίος θα παρουσιάσει τους ε, ομιλητές Ήθελα να ξεκινήσω την εδρίαση με μερικά σχόλια. Βασικά, να σας πω ότι είναι η τελευταία ακρόαση της Επιτροπής σε αυτή τη θητεία. Καλό που επιλέξαμε το θέμα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε επεξεργαστεί πολύ. Κατά τη διάρκεια της θητείας μας είχαμε σημαντικές εκδηλώσεις ανθρωπιστική βοήθεια. Είχαμε την Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής για Ανθρωπιστική Βοήθεια Θέλαμε να δώσουμε νέο ορισμό για την ανθρωπιστική βοήθεια και ένα τρόπο εργασίας στον τομέα αυτό, στον 21ο αιώνα. Και είχαμε και μεγάλες κρίσεις τα τελευταία χρόνια που έπρεπε να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τους εταίρους της. Mm, Θα ήθελα λοιπόν να αποτίσω φόρο τιμή σε δύο ανθρώπους. Στον Επίτροπο τον κύριο Στυλιανίδη ήταν η τελευταία επίσημη συνάντηση μαζί μα στην Επιτροπή, διότι είναι δύο συνεδριάσει μα απομένουν πριν τι εκλογέ, κύριε Στυλιανίδη. Να αποτίσω φόρο τιμή στον κύριο Στυλιανίδη, διότι ήταν έξοχο Ευρωπαίο Επίτροπο την τελευταία πενταετία. Όλα ξεκίνησαν με τον Brexit. Όχι τον Brexit, όλο τον Brexit έχω στο μυαλό μου. Τελειώνει με τον Brexit. Όλα, όλα ξεκίνησαν με την έμπολα. Την κρίση της έμπολα όταν πρώτο αναλάβα τα καθήκοντα σαν επίτροπο και γινόταν, νίκατε συντονιστή Ευρωπαϊκή Ενώσεω για το έμπολα, τον ιό τη έμπολα. Μετά είχαμε την κρίση των προσφύγων από τη Συρία, την κρίση στη Συρία, τη συγκρούση στη Συρία. Δεν θέλω να την αποκαλώ κρίση, διότι όπω λέει η Φεντερίκα Μογκερή, ήταν κρίση για αυτού και όχι για μα. Εργαστήκατε πολύ σκληρά για να βελτιωθεί η υποδοχή των προσφύγων στην Ευρώπη. Εργαστήκατε επίσης πολύ σκληρά, ώστε να δοθεί αποστήριξη ανθρωπιστική σε χώρε όπω η Ελλάδα που είναι στην πρώτη γραμμή που έπρεπε να αντιμετωπίσει η Ελλάδα το θέμα των προσφύγων. Είχαμε το Μιανμάρ, μετά Νότιο Σουδάν, Βόρεια Νιγηρία, πρόσφατα τη Βενεζουέλα. Πάντα ήσασταν εκεί, πάντα πηγαίνατε επί τόπου, όπου υπήρχε κρίση. Είπατε ότι είσαστε κουρασμένο, δεν με εκπλήσει. Έχετε πάντα φορτωμένο πρόγραμμα και σήμερα φεύγετε. Θα πετάξετε τα πάτε σε άλλη συνεδρίαση. Θα πρέπει να φύγετε νωρί από την ακρόαση. Ευχαριστώ σε εσά να καταγραφεί τα πρακτικά τη συνεδριάσεω ότι σας ευχαριστούμε για ό,τι κάνατε. Θα τα ξαναπούμε, το ξέρω, πριν το τέλος της θητείας της κοινοβουλευτικής, αλλά επίσημα ήθελα να καταγραφεί αυτή η ευχαριστία, να ευχαριστήσω και τον Ρίκο Γκερέρο Σαλόμ, που ήταν μόνιμος ε, εισηγητής μας για την ανθρωπιστική βοήθεια και που ε, έφθετε πολύ, τα, υποσημείωνε πρακτικά προβλήματα στην Επιτροπή και προσφεύγουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το μετωπίσουμε. Είδαμε αυτό τον γκόμβο, τη διασύνδεση υπάρχει μεταξύ ανθρωπιστική βοήθειας και αναπτυξιακή βοήθειας. Βλέπουμε επιτόπου τον κόσμο που ζει επί πάρα πολλά χρόνια σε καταβλισμούς προσφύγων έκανε πολλή δουλειά με τον Επίτροπο Ενρίκε μαζί με τον Επίτροπο για την παιδεία και αυτό είναι μεγάλο ε, επίτευγμα. εξοδεύουν πολλά, πολύ περισσότερα χρήματα για την εκπαίδευση των παιδιών στα πλαίσια τη προσφυγική κρίση. Αυτό δεν το σκέφτεται πολύ συχνά ο κόσμο εκτό του πλαισίου. Εγώ δεν το είχα σκεφτεί. Μέχρι όταν ένα νέο στην εκλογική μου περιφέρεια μου είπε, ήταν από τη Σομαλία και πέρασε 11 χρόνια τη ζωή του σε καταβλισμό προσφύγων στην Κένια. Και μου είπε ότι έχασε όλη του την εκπαίδευση. Διότι σε αυτό το στατόπεδο, στον καταβλισμό τότε, δεν υπήρχε πρόβλεψη για εκπαίδευση. Μπόρεσε να καλύψει το, αυτή την υστέρηση. Όταν βρήκε μια θέση στο Ηνωμένο Βασίλειο τελικά σαν πρόσφυγας, έγινε δεκτός σαν πρόσφυγας, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για τους νέους ε, για να έχουν παιδεία. Κάντε τεράστια δουλειά και στι επιτροπέ. Και εσείς συγηθήκατε Ρίκε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χωρίς να χρονοτριβήσω, θα καθίσω εκεί να ακούσω τις ε, παρουσιάσεις και να δώσω το λόγο στον Ενρίκε που θα προεδρεύσει Να χειροκροτήσουμε τον Επίτροπο και τον Ρίκε Γκερέρο για τη δουλειά που έχουν κάνει. Θα μιλήσω ισπανικά. Γι' αυτό, όσοι χρειάζεστε, να βάλετε τα ακουστικά σας, παρακαλώ. Και θα πω δύο λόγια στα αγγλικά για το Χρήστο Στελιανίδη μόνο. Όντως, είμαστε συνάδελφοι, φίλοι και άνθρωποι που έχουμε αναλάβει ανά τον κόσμο δεσμεύσεις για τα θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας. Όπως είπε και η Λίντα Μαγκάβαν, σας θεωρούμε όχι ως επίτροπο, αλλά ως φίλο, ως κάποιο με τον οποίο συνεργαστήκαμε τα πέντε τελευταία χρόνια και θυμάμαι τις δύσκολες στιγμές που ήταν ε, τα πρώτα τα πρώτα hearings που είχαν γίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για σας πριν να λάβετε. Και καταλαβαίνετε πόσο σημαντική και συγκινησιακή μετά από τόσα χρόνια είναι η σχέση μας. Σε ευχαριστούμε πολύ Χρήστο, έχεις το λόγο. I'm feel little bit shy, Κάπως ε, ντροπαλός αισθάνομαι με αυτά που άκουσα. Τα, όλα αυτά τα ευγενικά λόγια από τους αγαπημένους συναδέλφους, τη Λίντα και τον και Στην προηγούμενη συνεδρίαση εξέφρασα όχι μόνο τη βαθιά μου εκτίμηση για την συνεργασία που έχω με την Επιτροπή Ανάπτυξης, αλλά κυρίως για τη φιλία που αναπτύξαμε. Και όπως είπαν ήδη και ο Ενρίκε και η Λίντα, αρχίσαμε ως συνάδελφοι. Κατά τη διάρκεια αυτή τη τόσο δύσκολη περίοδου, κατά τη διάρκεια τη οποία αντιμετωπίσαμε σοβαρά προβλήματα. Την έμπολα, διάφορες ε, κρίσεις, την προσφυγική κρίση. Αλλά στην πρώτη φάση της συνεργασίας μας κατορθώσαμε να γίνουμε φίλοι διότι συμμεριζόμαστε στις αρχές και τις αξίες. Σας ευχαριστώ λοιπόν και είμαι σίγουρος ότι στην Επιτροπή Ανάπτυξης χωρίς τη Λίντα ως ε, ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα χάσουμε πολλά πράγματα και εμείς και ο Ενρίκε είμαστε ε, πάρα πολύ φανατικοί για όλα αυτά τα θέματα το, σε τις βοήθειες και όλα τα άλλα με τα οποία θα... Χάρη στη Λίντα. Ε, είναι σαφές αυτό που λέτε, ναι, ναι, ναι. Συγχρόνως όμως, θα πρέπει να πω ότι ελπίζω ότι και πάλι θα ξαναδώ τον Ενρίκε στην ε, νέα θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί έχουμε ανάγκη από την σοφία που διαθέτεις, Ενρίκε. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά πρόκειται για μια μεγάλη πρωτοβουλία. Το θέμα που θα συζητήσουμε, δηλαδή το μέλλον της ανθρωπιστικής βοήθειας, το οποίο είναι απόδειξη των κοινών δεσμεύσεων που έχουμε αναλάβει και ιδιαίτερος για να μελετήσουμε τους τρόπους με τους οποίους θα βοηθήσουμε περισσότερους ανθρώπους και με καλύτερο τρόπο. Αγαπητοί φίλοι, και απευθύνομαι ιδιαίτερα στα άτομα τα οποία βρίσκονται εδώ στην έδρα μαζί μας. Ξέρουν ποιες είναι οι δυσκολίες, ακόμη καλύτερα και από εμάς. Υπάρχουν 132 εκατομμύρια άνθρωποι που χρειάζονται την ανθρωπική βοήθεια το 2019. 69 Σε 69 εκατομμύρια ανέρχεται η βοήθεια. Η Ουγγάντα, ο το Μπαγκλαντές, το Σουδάν και η Τουρκία μοιράζονται 85% του βάρους των ε, μετακινηθέντων ατόμων. Δεν είναι οι μόνες χώρες όμως. Η κλιματική αλλαγή, οι φυσικές καταστροφές είναι όλο και περισσότερο αιτίες θανάτου και καταστροφικών όρων διαμονής και αναγκαστικής μετακίνησης εκατομμυρίων ανθρώπων. Η μέση ανθρωπιστική κρίση σήμερα διαρκεί περισσότερο από 9 χρόνια. Και οι έκτακτε καταστάσει που δημιουργούνται δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν παράδοξο για όλου. Πριν από 10 χρόνια, ίσω αυτού του είδου η ορολογία ήταν κάτι που δεν χρησιμοποιείται συχνά. Σήμερα όμω πρόκειται για μια κατάσταση η οποία έχει. Ε, πρόκειται για εκφράσει που θεωρούνται κοινέ. Και βεβαίω ξέρουμε ότι ξεπερνώνται οι δυνατότητε που διαθέτουμε. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώ θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη νέα σκληρή πραγματικότητα και για τον τρόπο αυτό στην τελευταία ανταλλαγή απόψεων που είχαμε πριν από μερικές εβδομάδες, επέμεινα σε ένα θέμα. Είπα ότι το πώς προσφέρουμε, παραδίδουμε και την ανθρωπική βοήθεια είναι τόσο σημαντικό όσο την ίδια την αρχή αυτής. Γι' αυτό θα πρέπει να εστιάσουμε σε αυτό το θέμα την προσοχή μας, ώστε να ενεργήσουμε με πιο αποτελεσματικό, καινοτόμο και βεβαίως πιο βιώσιμο τρόπο. Επιτρέψτε μου να πω για αυτά τα τρία θέματα που προανέφερα να πω κάτι, διότι από την εμπειρία μου στον τομέα αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να βαθύνουμε τη συζήτηση. Πρώτα απ' όλα, η καινοτομία. Όταν μιλώ για καινοτομία, σκέπτομαι το συστήματα ε, χορήγησης voucher και ε, ρευστού. Πρόκειται για ένα ευέλικτο σύστημα που δίδει στα ευάλωτα άτομα την δυνατότητα να αντιμετωπίζουν τις καθημερινές τους ανάγκες αξιοπρεπώς, ανεξάρτητα και με αξιόπιστο τρόπο. Αυτό είναι κάτι το οποίο αυξάνει και την αποτελεσματικότητα, μειώνει τα γενικά έξοδα, αυξάνει την πραγματική, την καθαρή αξία της βοήθειάς μας και προσφέρουμε περισσότερα με λιγότερο δαπανηρό τρόπο. Είδα εξαιρετικά αποτελέσματα σε πολλές χώρες. Πολλοί από εσά γνωρίζετε το ESSN στην Ιορδανία, στο Λίβανο και ακόμη και στην Ελλάδα. Υπήρχαν κάποιες καθυστερήσεις μέχρι να μπορέσουμε να θέσουμε σε εφαρμογή αυτή την εξαιρετική διαδικασία, αλλά όταν το κατορθώσαμε, πραγματικά είδα ότι οι Σύριοι πρόσφυγες αισθάνθηκαν πολύ καλύτερα διότι απέκτησαν ε, ε, αξιοπιστία και αισθάνθηκαν ότι μπορούν με αξιοπρεπή τρόπο να αντιποκριθούν σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες ζωής. Παραδείγματος χάρη, το 2017 περίπου 4% του συνολικού ποσού ε, δόθηκε μέσω cash και voucher. 900 εκατομμύρια δολάρια. 4% είναι μεγάλο ποσό. Αρχίσαμε από το 2011. Το 2018 συνεχίστηκε αυτή η τάση και βεβαίως θα συνεχιστεί και φέτος. Πρόκειται για το ανώτατο ρεκόρ το οποίο έχουμε φτάσει στα πλαίσια της ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε, χρειαζόμαστε λοιπόν και τη συνδρομή σας, τη βοήθειά σας για να μπορέσουμε αυτό το αποτελεσματικό αλλά απαιτητικό μέρος της βοήθειας να μπορέσουμε να το συνεχίσουμε και το φέρουμε σε πέρας με επιτυχία. Επιτρέψτε μου τώρα να αναφέρω κάποια πολύ σημαντικά παραδείγματα. Στην Ιορδανία έχουμε τεχνολογία αναγνώρισης ε, για να καταγράφουμε τους πρόσφυγες. Στην Τουρκία δίδεται ε, μεγάλο ποσό για να μπορέσει να υπάρχει για κάθε άτομο μία ενιαία ε, πιστοτική κάρτα που να μπορεί να δίνει ρευστό και βεβαίως ε, χρειάζεται και η κατάλληλη εκπαίδευση των ατόμων που χειρίζονται αυτά τα θέματα. Χρειάζεται ένας αποτελεσματικός τρόπος για να μπορέσουν να πολλαπλασιαστούν οι δυνατότητες ε, για τα παιδιά να βοηθηθούν και να πάνε στο σχολείο. Στη Σομαλία επίσης. Δόθηκε ρευστό μέσω των ε, διαφόρων εταιριών κινητή. Στην ε, ε, Ελλάδα θεσπίσαμε το πρόβλημα εστία και δώσαμε ε, ήδη προπληρωμένες κάρτες στους πρόσφυγες και μετανάστες για να καλύψουν τις ανάγκες τους και είναι αυτό το πράγμα και υποφελές για τις διάφορες τοπικές αγορές. Θα ήθελα να πω εδώ το εξής. Όταν επισκέφθηκα το Καζιαντέπ είχα μια πολύ καλή εμπειρία. Πριν να πάω στο Gaziantep, είχαμε πολλά προβλήματα μεταξύ των κοινοτήτων υποδοχής και των προσφύγων, κυρίως στην ε, αρχή όπου υπήρχαν πάρα πολλά άτομα που ερχόντουσαν ε, από διάφορες περιοχές της Συρίας. Το Χαλέπι κι άλλες. Όταν λοιπόν έφτασα εκεί είδα ότι η τοπική οικονομία και η τοπικοί επιχειρηματίες ε, υποφελούνταν από αυτά τα cash and vouchers και είδα ότι μέσω αυτού του μέσου μπορέσαμε και να ε, ξαναδώσουμε πίσω την αξιοπρέπειά τους στους πρόσφυγες, αλλά δημιουργήσαν και καλύτερες συνθήκες συνύπαρξης μεταξύ των κοινοτήτων υποδοχής και των κοινοτήτων των προσφύγων. Και πραγματικά υπήρχε αυτό το συνέστημα, το θετικό επιτόπου το διαπιστώσαμε κι εμείς. Ξέρω ότι δεν έχω πολύ χρόνο, περνώ στο δεύτερο θέμα μου. Όλοι μας μιλούμε πάντα για αποτελεσματικότητα. Ε, but uh, what does... Είναι μαγική η λέξη αυτή, αλλά τι σημαίνει ο όρος αποτελεσματικότητα. Σημαίνει πρώτα και κύρια καλύτερη αξιοποίηση των υπαρχόντων δημοσιονομικών σπόρων. Αξιοποίηση καλύτερη της ανθρωπιστικής μας βοήθειας. Γιατί κάθε ευρώ που δαπανούμε μετατρέπεται σε ένα ευρώ το οποίο βοηθά ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια. Γίνεται φαγητό, γίνεται κουβέρτες, γίνεται εμβόλια και με αυτόν τον τρόπο στις διαπραγματεύσεις μας, στις διαβουλεύσεις μας με τους εταίρους μας επιμένουμε πάντοτε σε αυτή την πτυχή, διότι πάνω απ' όλα έχουμε καθήκον να προστατεύσουμε τους ε, οικονομικούς μας πόρους βεβαίως, αλλά ταυτόχρονα, και αυτό είναι πολιτικό ζήτημα, και δυστυχώς οι ευρωβουλευτές γνωρίζετε πολύ καλά ότι Ιδίω κάποιοι άνθρωποι και εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο αλλά και στα Εθνικά Κοινοβούλια προσπαθούν να καταστρέψουν τη φήμη της αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας υπερβάλλοντας όσον αφορά τις παροχές που δίνονται. Πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό το πρόβλημα για να έχουμε καλά επιχειρήματα ε, απέναντι σε εκείνους που ισχυρίζονται ότι η αναπτυξιακή και ανθρωπιστική βοήθεια δεν είναι απαραίτητη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για μας αυτό δεν είναι απλώς μια υποχρέωση, είναι ηθικό καθήκον μας. Πρέπει να κερδίσουμε αυτή τη συζήτηση για να μπορέσουμε να αποκρούσουμε αυτήν την λαϊκιστική τροπή που έχει πάρει πολλές φορές η συζήτηση. Να επιμείνουμε στη σημασία που έχει η ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα. Στην Ελλάδα, μέσα από την συμφωνία μας με την ύπατη αρμοσία, αναπτύξαμε, αυξήσαμε μάλλον το κόστος της παροχής σε πάνω από 5%. Είναι εντυπωσιακή, ε, εντυπωσιακό αυτό το αποτέλεσμα. Στην Τουρκία όλα τα προγράμματα έχουν ε, ποσοστό 6,5% έμεσου κόστους που είναι ακριβώς το ίδιο ποσοστό που έχουμε, συμφωνήσει και στις, που έχουμε καθορίσει και στις με τον Ερυθρό Σταυρό. Και ξέρετε, εγώ το χρησιμοποιώ αυτό το επιχείρημα πολύ συχνά στις ε, επαφές μου με κυβερνήσεις των κρατών μελών και πραγματικά είναι πάρα πάρα πολύ ισχυρό το επιχείρημα αυτό όταν θέλει κανείς να αντικρούσει εκείνους που αντιτίθενται στην έννοια της ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας. Δεύτερο σημείο. Αποτελεσματικότητα σημαίνει και καλύτερη αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων. Η πραγματοποίηση επενδύσεων σε τοπικές εταιρικέ σχέσεις ήταν μία από τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε το 2016 στη Διεθνή Διάσκεψη για την Ανθρωπιστική Βοήθεια που έγινε στην Κωνσταντινούπολη. Πιστεύουμε πολύ στο να γίνουν επενδύσεις στις δυνατότητες και στις γνώσεις των τοπικών μας εταίρων. Ταυτόχρονα η ανθρωπιστική βοήθεια, η αναπτυξιακή βοήθεια θα πρέπει να υπόκειται σε διαφανή διαχείριση. Εμείς βοηθούμε, υποστηρίζουμε τους τοπικούς εταίρους μας, τους βοηθούμε να διαχειρίζονται με τη δέουσα επιμέλεια τα κονδύλια που λαμβάνουν και τους βοηθούμε να αναπτύξουν τις δικές τους ικανότητες. Γιατί περισσότερο από το να δίνει κανείς χρήματα είναι πολύ σημαντικό να βοηθήσει τους εταίρους του επιτόπου να μπορούν οι ίδιοι να επιτυχάνουν τους στόχους. Και ξέρετε κι εσείς όλοι σας πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των τοπικών εταίρων μας. Εγώ αποκόμισα πάρα πολλές εμπειρίες στις επιθέσεις της Μποκοχαράμ, στην Ιορδανία, στο Λίβανο και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι οι τοπικοί εταίροι μας ξέρουν καλύτερα από εμάς, ξέρουν τις τοπικές περιστάσεις, το περιβάλλον και μπορούν πολύ καλύτερα να χειρίζονται και να προσεγγίζουν τα θέματα τα προβλήματα από ότι εμείς που είμαστε απ' έξω. Χθες έγινε μια συνδιάσκεψη στη Γενέβη για την Ιεμένη. Και εγώ συμμετείχα σε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση για την ψυχική υγεία με τον ε, Πίτερ Μάουελ, τον ε, Υπουργό Ανάπτυξη των Κάτω Χωρών. Και συνειδητοποίησα, και αυτό ήταν πολύ σημαντικό για μένα, παρά το γεγονός ότι είμαι γιατρός, ότι κάποιες φορές οι τοπικοί εταίροι μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για να αντιμετωπιστούν και τα προβλήματα ψυχικής υγείας επιτόπου. Και οι τοπικοί εταίροι ακριβώς αυτό τόνιζαν. Αλλά και η ευρωπαϊκή πλευρά. Τόνιζαν όλοι πόσο σημαντικό είναι να έχει κανείς τοπικούς εταίρους ώστε να μπορούν εκείνοι να αναλαμβάνουν την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση διαφόρων ε, προβλημάτων. Ξέρω, δεν έχουμε χρόνο. Θέλω μόνο να πω κάτι για την βιώσιμη ευρωπαϊκή ανθρωπιστική βοήθεια. Γνωρίζετε ότι η παιδεία συνδέεται εξορισμού με το μέλλον. Προσφέρει ανθεκτικότητα, βιωσιμότητα, εξασφαλίζει την ειρήνη. Και γι' αυτό το λόγο τονίζω και επικεντρώνομαι πάντοτε στην, στο θέμα της παιδείας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για εμένα. Το 2019, φέτος, ανταποκρινόμαστε στη δέσμευσή μας να δοθεί το 10% της ανθρωπιστικής μας βοήθεια σε εκπαίδευση και κατάρτιση, από την πρόσβαση στην ε, παιδεία έως και την ε, βελτίωση της ποιότητας της ε, παιδείας και από τον Μάιο έχουμε θέσει σε εφαρμογή και το πρώτο πλαίσιο πολιτικής για την παιδεία ε, σε ε, εμπόλεμες ζώνες με την απαραίτητη υποστήριξη και της δικής σας Επιτροπής, της Επιτροπής Ανάπτυξης, γιατί ήταν πάρα πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε τη δική σας υποστήριξη προκειμένου να περάσουμε αυτό το 10% του προϋπολογισμού και να κατευθυνθεί στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Συνάδελφοι, λοιπόν, θα έλεγα ότι έχουμε επιτύχει αρκετά πράγματα, όμως μένουν και πολλά ακόμη να γίνουν. Να μην ξεχνάμε ότι η ανθρωπιστική βοήθεια βεβαίως δεν μπορεί από μόνη της να δώσει την απάντηση στην, στον εύσταυτο χαρακτήρα σε πολλές κρίσεις. Φυσικά χρειάζονται συντονισμένες λύσεις ολοκληρωμένες λύσεις, ολοκληρωμένε απαντήσεις οι οποίες θα περιλαμβάνουν την αναπτυξιακή, την ανθρωπιστική βοήθεια και ε, τις ειρηνευτικέ προσπάθειες. Μια σύνδεση των τριών αυτών ενιών η οποία σε καμία περίπτωση δεν θα υποσκάπτει τις βασικές μας αξίε. Και επιμένω σε αυτό γιατί κάποιε φορές υπάρχουν συνομιλητέ μας οι οποίοι θεωρούν ότι αυτή, αυτή, αυτό το τρίπτυχο θα μπορούσε να καταστρέψει ακόμα και τις αρχές μας για την ανθρωπιστική βοήθεια. Όχι, σε καμία περίπτωση δεν καταστρέφει, δεν, καταστρέφει, δεν, δεν παραβιάζει τις αρχές μας. Πρέπει απλώς να είμαστε αποτελεσματικοί και να σας πω την αλήθεια αυτό το τρίπτυχο αυτή η διασύνδεση των τριών πτυχών που σας ε, παρουσίασα μπορεί να εφαρμοστεί μόνο αν υπάρχουν πραγματικά εφικτές λύσεις που θα αποβαίνουν προς όφελος των ανθρώπων που πλήττονται από τις κρίσεις. Και για να γίνουν όλα αυτά χρειάζεται να έχουμε μια πολύ ευρύτερη και ολοκληρωμένη εικόνα για τα ριζικά αίτια των κρίσεων. Πρέπει να έχουμε εργαλεία για τον μετριασμό των καταστροφών, την αντιμετώπιση των κρίσεων και χρειαζόμαστε για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός πολιτικούς συμμάχους. Αυτή η προσέγγιση της διασύνδεσης λοιπόν ήδη αποφέρει αποτέλεσμα στις έξι πιλωτικές χώρες όπου εφαρμόζεται. Σουδάν, στο Σουδάν έχουμε καταφέρει και έχουμε μειώσει σημαντικά τα ποσοστά του υποσυτισμού κατευθύνοντας εργαζόμενους στα συστήματα κοινωνικής προστασίας. Με τις δράσεις μας στην Ουγκάντα καταφέραμε και εντοπίσαμε έγκαιρα τις ροές των ε, προσφύγων και το πού κατευθύνονταν. Έχουμε λοιπόν απτά αληθινά παραδείγματα του πώς η ανθρωπιστική βοήθεια μπόρεσε να βοηθήσει μέσα από αυτή την διασύνδεση των ε, τριών πτυχών που σας ανέφερα. Η ανθρωπιστική βοήθεια λοιπόν ε, έχει ως στόχο της να απαλύνει τον πόνο και τα βάσανα των ανθρώπων που πλήττονται από τον πόλεμο, τη φτώχεια, την κλιματική αλλαγή. Χρειάζεται λοιπόν να παρέχεται με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Θα συμμετάσχω στην έκτη παγκόσμια ε, πλατφόρμα για την μείωση των ε, αρνητικών επιπτώσεων των κρίσεων που θα γίνει το Μάιο στην Γενέβη. Και θέλω πραγματικά το έργο μας εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτελέσει σημείο αναφοράς των συζητήσεων. Αντίστοιχες συζητήσεις, ξέρετε, είχαμε κάνει και στο παρελθόν και στο Κανκούν και νομίζω ότι αγωνιστήκαμε σκληρά για να, για να πείσουμε και τις άλλες αντιπροσωπείες ώστε να κατανοήσουν την αναγκαιότητα του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πόσο σημαντικό είναι να λαμβάνεται υπόψη και η Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, διότι αυτά είναι θέματα που συμβαδίζουν. Να ολοκληρώσω. Η ανθρωπιστική βοήθεια που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση προφανώ δεν μπορεί να αποτελέσει πανάκια και να επιλύσει όλα τα προβλήματα και τι προκλήσει που αντιμετωπίζει ο κόσμο μα. Ούτε μπορεί να επιλύσει όλα τα πολιτικά προβλήματα. Όμω, η ανθρωπιστική βοήθεια που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απαραίτητη, είναι αναγκαία και από τι εμπειρίες μα έχει αποδειχθεί ότι είμαστε ένα αξιόπιστο παγκόσμιο εταίρος, εταίρος με συγκεκριμένε αξίε και προτεραιότητες. Ο νέος πρωθυπουργός της Αιθιοπίας και ο νέος πρωθυπουργός της Ιεμένης χθες μου είπαν αμφότεροι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο πιο αξιόπιστος εταίρος τους. Και να σας πω την αλήθεια, ένιωσα περήφανος για τη βοήθεια που έχουμε παράσχει και στην Ιεμένη και στην Αιθιοπία. Και είναι μια μορφή αναγνώρισης το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο πιο αξιόπιστος εταίρος τους. Και έτσι μπορούμε να πούμε και στους πολίτες μας ότι μπορούμε να συνεχίσουμε και να αυξήσουμε την ανθρωπιστική βοήθεια που χορηγούμε. Και γι' αυτό το λόγο, μέσω του σώματος των επιτρόπων, έχουμε προτείνει 30% αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Έχει λοιπόν δημιουργηθεί μια σημαντική δυναμική για την ανθρωπιστική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειαζόμαστε πραγματικές λύσεις, πρακτικές λύσεις για πραγματικούς ανθρώπους. Είναι καιρός να σκεφτούμε με τρόπο καινοτόμο να αξιοποιήσουμε νέα εργαλεία όπως το Cash and Voucher, να εμπλέξουμε νέους φορείς, ιδίως τοπικούς, για να συνάψουμε εταιρικέ σχέσεις με άλλες χώρες γειτονικέ όπως έχουμε κάνει και στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Και θέλω να πω μία κουβέντα ακόμη. Χρειαζόμαστε και τον ιδιωτικό τομέα. Πρέπει να βρούμε τρόπους να πείσουμε τον ιδιωτικό τομέα ότι το, θέμα, το πρόβλημα, τα προβλήματα μας αφορούν όλους. Συνάδελφοι, όπως είπα, είμαι πολύ περήφανο για όλα όσα καταφέραμε τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Είμαι βαθιά πεπισμένο ότι μπορούμε να κάνουμε ακόμη περισσότερα πράγματα υπέρ εκείνων που χρειάζονται πιο πολύ από όλου την βοήθειά μας. Είναι ευθύνη μα και καθήκον μας για την ε, ευρωπαϊκή μας ταυτότητα. Γιατί έχω πει πολλές φορές ότι η αρχή της ανθρωπιστικής βοήθειας αποτελεί εγγενές τμήμα της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Αποτελεί τμήμα των ηθικών μας υποχρεώσεων. Ευχαριστώ. Now it's true that Αληθεύει. Πράγματι θα μιλήσω σπανικά τώρα πια. Όχι όπως έκανα πριν. Κύριο Ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για την παρέμβασή του και κατά κάποιον τρόπο πρόκειται για τον απολογισμό που κάνει μετά από πέντε χρόνια στην θέση αυτή. Πρόκειται απολογισμό για το τι κάναμε, αλλά και για επιβεβαίωση των δεσμεύσεων που έχουμε λάβει για το μέλλον. Σε λίγους μήνες, όπως ξέρουμε, θα γίνουν εκλογές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα έχουμε ένα νέο διαφορετικό κοινοβούλιο μετά, αλλά όλοι θα πρέπει να προσπαθήσουμε ώστε να γίνει πραγματικότητα η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το κονδύλι ε, για την ε, ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει τα 11 δις, ώστε, όπως είπε και ο Επίτροπος, να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Όντω, κάποιοι από εμά δεν θα είναι πλέον εδώ. Υπάρχει ζωή και εκτό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το ξέρουμε, αλλά αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αγωνιζόμαστε, είναι να υπάρχει και ζωή μετά από κάποια ανθρωπιστική κρίση. Μετά από ένα, μια φυσική καταστροφή, μετά από κάποιο πόλεμο. Νομίζω ότι αυτή πρέπει να είναι η μεγάλη δέσμευσή μας και δέσμευση την οποία πρέπει να περάσουμε και στην επόμενη ε, μη των συναδέλφων εδώ και ο Χρήστος στην επόμενη ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, επειδή έχει και άλλες υποχρεώσεις, ο κύριος Επίτροπος θα πρέπει να φύγει. Αν θέλει κάποιος να κάνει τώρα μία μικρή παρέμβαση, να κάνει μια ερώτηση, του δίνω μέσα στο λόγο. Νόρμπερτ. Äh, Ευχαριστώ πολύ τον Επίτροπο για αυτά που μας είπε. Και ευχαριστώ και τον Ενρίκε, τον ε, μόνιμο εισηγητή μας για τα θέματα αυτά. Νομίζω ότι ε, όλος, το όλο σχήμα ήταν πάρα πολύ ευτυχές και πετυχημένο. Ε, είχαμε τον κύριο Στυλιανίδη, τον Επίτροπο και τον Ερή και τον μόνιμο εισηγητή μας και τη Λίντα Πρόεδρο της Επιτροπής ε, Ανάπτυξης και θέλω να υπογραμμίσω ότι η χημεία πάντα ήταν υπέροχη, έξοχη και σε όλη την Επιτροπή. Και με υπερηφάνεια μπορεί να λέει ο κύριος Επίτροπος ότι όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια έχουμε συνεργαστεί άριστα. Εάν στο τέλος της ε, υπάρχουν ερωτηματικά σχετικά με την πρόοδο που επετεύχθη. Μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πετύχει πρόοδο. Η ανθρωπιστική βοήθεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο πραγματικά έχει γίνει πιο πιστική. Αν μας πούνε αν ήμασταν καινοτόμοι, ήμασταν καινοτόμοι, γίναμε πιο πιστικοί, γίναμε καινοτόμοι μέσω νέων τεχνικών που χρησιμοποιήθηκαν, όπως έδειξαν κατά διάφορα παραδείγματα που παρετέθησαν. Και θέλουμε να στηρίξουμε την αξιοπρέπεια των προσφύγων. Και τελικά ανταποκριθήκαμε και σε ευθύνε μα, πιστεύω. Μπορώ, αν μα ρωτήσουν αυτό, αν ανταποκριθήκαμε στι ευθύνε μα, μπορούμε να πούμε ναι. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τις ΜΚΟ και τις διάφορες, ε, φορεί φορείς του οργανισμού οργανισμούς που παρήχαν βοήθεια, του οργανισμούς συνδρομής. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ήταν εξαιρετική εταίρη. Αλλά αυτό που απομένει μετά τη θητεία και πώς θα εξελιχθούν περαιτέρω τα πράγματα είναι το θέμα. Αν δείτε το όλο σχήμα, τον αστερισμό, το ΣΥΠΗΝ που ίσως σχηματιστεί μετά τις εκλογές, ίσως τελικά τότε είναι μικρότερη οικογένεια που κινήθηκε προς τη σωστή κατεύθυνση ανθρωπιστική βοήθεια. Ίσως υπάρχουν αντιστάσεις από περιοχές, από χώρους που υπάρχει μικρότερη αλληλεγγύη και επικρατεί περισσότερο εγωισμός και η πολυμερής προσέγγιση ίσως να μην λαμβάνεται υπόψη τόσο πολύ και οι διάφορες κοινέ αξίες της Ευρώπης ίσως να αμφισβητούνται, ίσως αλλάξουν τα πράγματα. Άρα θα πρέπει να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα αν προκύψουν. Και νομίζω ότι αυξάνοντας τους πόρους που διατίθενται, τα χρήματα που διατίθενται, στείλαμε ένα αποφασιστικό ξεκάθαρο μήνυμα. Και χαίρομαι όλος ιδιαίτερος επίσης και είμαι ευγνώμων, διότι μέσω του Ενρίκε ο ρόλος της ανθρωπιστικής ε, βοηθείας τονίστηκε. Χωρίς βιωσιμότητα όμως αυτής της βοήθειας, χωρίς μελλοντικές προπτικές, νομίζω ότι θα ακολουθούσαμε λάθος προσέγγιση. Από την πλευρά μου και από πλευρά της πολιτικής μου ομάδας θα ήθελα ξανά να ευχαριστήσω όλους που συμμετείχαν στην προσπάθεια. Ήταν δύσκολα τα χρόνια που περάσαμε με πάρα πολλά προβλήματα και προκλήσεις, αλλά γενικά πρέπει να πω ότι νομίζω ότι κάναμε αρκετά καλή δουλειά, συλλογική δουλειά και μετά τις εκλογές με τα χαρά θα ήθελα να εργάζομαι σε αυτόν τον τομέα και ελπίζω ότι οι προαναφερθέντες συντελεστές θα συνεχίσουν και μετά τις εκλογές να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους και να συνεχίζουν να ε, προωθούν την ανθρωπιστική βοήθεια, να επεξεργάζονται το θέμα τη ανθρωπιστική βοήθεια. Και θα είναι πολύ καλύτερο για την ανθρωπιστική βοήθεια αν παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τελικά το Ηνωμένο Βασίλειο. το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Στυλιανίδη Και εγώ εκ μέρους των Πρασίνων θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία που είχαμε. Ε, ήταν πραγματικά πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι ήσασταν πάντοτε πρόθυμος να μας ακούσετε. Από, τις, από τα όσα μας είπατε, βλέπω ότι δεν σας ενδιαφέρει μόνο η παροχή της ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά πώς θα συνεχίσουν τα πράγματα στη χώρα που κάθε φορά λαμβάνει την ανθρωπιστική βοήθεια και ιδίως αυτό που αναφέρατε για τα cash and vouchers ε, για την τόνωση και της τοπικής οικονομίας είναι πραγματικά ε, ήταν μια εξαιρετική ιδέα είναι μια εξαιρετική ιδέα. Ίσως θα μπορούσαμε να βασιστούμε σε αυτή την ιδέα και να την ε, αναπτύξουμε περαιτέρω. Γιατί νομίζω ότι όταν εξασφαλίζεται η συμβίωση των ανθρώπων και για τη συμβίωση βεβαίως ε, είναι μια προϋπόθεση και η οικονομική δραστηριότητα, τότε μπορούν στην πράξη να λύνονται προβλήματα. Εγώ προσωπικά δυστυχώς δεν θα είμαι στη νέα θητεία του Κοινοβουλίου. Ελπίζω όμως τα νέα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συνεχίσουν με την ίδια ζέση, με την ίδια ε, θέρμη ε, το έργο που έχουμε αναλάβει Ιδίω ε, για, για τα θέματα της ανθρωπιστικής βοήθειας που κατευθύνεται προς την παιδεία. Με σοκάρατε με αυτό που είπατε. Τόσο πολλά χρόνια, 9 χρόνια βρέθηκε παιδί έξω από την εκπαίδευση. Μιλάμε για τεράστιο χρονικό διάστημα, είναι τραγωδία που με τη σειρά του βεβαίως αυτό μας δείχνει και πόσο σημαντική είναι αυτή η ανθρωπιστική βοήθεια να φτάνει στον προορισμό της έγκαιρα. Ε, ελπίζω λοιπόν και το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην ε, γλιστρήσει σε επικίνδυνες ατραπούς ε, ιδεολογικές και να συνεχίσει να προάγει την ανθρωπιστική βοήθεια που άλλωστε είναι και μια χριστιανική αξία. Σας ευχαριστούμε για όλα και ελπίζω να συνεχιστεί το έργο σας. Εκτός μικροφώνου ο Πρόεδρος. Το μικρόφωνο παρακαλούμε. Ο δεύτερος προσκεκλημένος μας είναι ο Ραβμπεφ Παφασίγκαν, διευθυντής του συντονισμού για την ε, επισητιστική βοήθεια Ότσο. Αυτή τη στιγμή είναι υπεύθυνο διαφόρων κλάδων της Ότσο και πριν ήταν συνσυντονιστής για τα θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ στη Συρία. Επίσης εργάστηκε στο Αφγανιστάν, στη Βοσνία Ζεγοβίνη, στην Παλαιστίνη, στο Σουδάν και έχει εμπειρία τουλάχιστον 25 ετών σε θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας. Έχετε το λόγο κύριε Ραμέσου. Uh, uh, uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, συγκεκριμένα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συνάδελφοι του πάνελ, κυρίες και κύριοι. Ξεκινώντας, θα πω ότι η Ευρώπη είναι ο μεγαλύτερος συνεισφορέας ανθρωπιστικής βοήθειας ανθρωπιστικά προγράμματα στον κόσμο. Χωρίς αυτή τη συνεισφορά εκατοντάδες χιλιάδες ζωές θα είχαν επηρεαστεί αρνητικά, ίσω να είχαν χαθεί, κυρίως η θνησιμότητα θα ήταν μεγαλύτερη και με μεγάλη ευγνωμοσύνη και εκτίμηση παριστάμεθα για να σε ευχαριστήσουμε για όλες τις προσπάθειές σας και την υποστήριξη προς τα προγράμματά μας. Να πω μερικά λόγια όσον αφορά το παγκόσμιο αυτό σύστημα ανθρωπιστικής βοήθειας. Τρία χρόνια πέρασαν από τη Σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη το 2016 και κάναμε βήματα στο, στον ΟΗΕ ε, έδωσε καρπούς. Αυτή η σύνοδος στην Κωνσταντινούπολη ήταν πολύ σημαντικό γεγονός, έθεσε στόχους πολύ φιλόδοξους. Η ανθρωπότητα θέτει καινούριου στόχους μέσω τοπικής και παγκόσμιας προσέγγισης ε, προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις ανθρωπιστικές ε, κρίσεις και θέλει να σταματήσει η ανθρωπιστική ε, βοήθεια μέσω της ανάπτυξης, να μην χρειάζεται πια. Ε, λοιπόν, η συνεργασία έχει συνεχιστεί στα ύψιστα επίπεδα, η αναπτυξιακή, και θα πρέπει να αναδημορφωθούν οι στατικές των κρατών μελών σε επίπεδο κρατών μελών. και τελικά εφαρμόζονται νέα μέθοδοι μετά από τη Σύνοδο Κορυφή. Υπάρχει έγκαιρη προειδοποίηση, ε, δραστηριοποιούνται νωρί τα κράτη-μέλη για να μειώνεται ο αντίκτυπο των κρίσεων. Έχουν τεθεί διάφορα νομικά και πλαίσια και πλαίσια πολιτική, άμεση χρηματοδότηση των τοπικών διοικήσεων για να επιτευχθούν συλλογικά αποτελέσματα. Εστιαζόμεθα περισσότερο στη ΣΟΤΑ και στα, κράτη, στα διάφορα κράτη για την απόξη της κρίσης και η διεθνής δράση πρέπει να γίνει πιο διαφανής, πιο αποτελεσματική, αποδοτική και ελεγχόμενη, κυρίως να μπορούν να βλέπουν πού πηγαίνουν τα χρήματα οι γενναιόδοροι δωρητέ. Αυτά τα βήματα έχουμε κάνει. Η πρόοδος ε, ήταν άνηση και περιοριζόταν η, τα επιτεύγματα στις υφιστάμενες δομές και λόγω των πόρων διότι οι ευάλωτοι άνθρωποι έχουν αυξηθεί σε πάρα πολύ σημαντικό βαθμό στον κόσμο. Για να πετύχουμε διθωτικές αλλαγές που θέλουμε, πρέπει να ξεπεράσουμε βραχυπρόθεσμες λύσεις και έχουμε μεγάλη ευκαιρία σήμερα ε, με τη διαδικασία μεταρρύθμισης που γίνεται στον ΟΗΕ να κινηθούμε από κοινού και να κάνουμε αυτό που είπε ο Επίτροπος κ. Στυλιανίδης, να φέρουμε την ανάκαμψη και να αποκατασταθεί αξιοπρέπεια των ανθρώπων τον ταχύτερο, το ταχύτερο δυνατόν τα προβλήματα ανθρωπιστικά παραμένουν ίδια. Ε, με σύγκρουση και σειράξεις ε, εστιάζεται τώρα σήμερα η δυστυχία των ανθρώπων. Παλιά ήταν οι φυσικές καταστροφές. Τώρα τα προβλήματα διαρκούν περισσότερα. Είναι πιο βία τα αποτελέσματα, πιο ομα... Και οι διάφορες ένοπλες ομάδες που συμμετέχουν σε ένοπλες σειράξεις έχει εκραγεί και είναι πολύ πιο δύσκολη η πρόσβαση πια και πολύ πιο δύσκολη η ρύθμιση των προβλημάτων. Και αυτό έχει συνέπειε ε, όσον αφορά την ασφάλεια και των φορέων που ε, δίνουν ανθρωπιστική βοήθεια. Χάσαμε εκατοντάδε εργαζόμενου στον τομέα ανθρωπιστική βοήθεια στη Συρία. Και έχουμε πάρα πολλού εκτοπιστέντε. Το είπε και ο Επίτροπο Στυλιανίδη. 70 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί λόγω των σειράξεων. Πολύ περισσότερο ποτέ κατά το παρελθόν. Σαν αποτέλεσμα αυτού, λάβοντα υπόψη αυτού του παράγοντε, έχουμε ετήσια ε, έχουμε τετραπλασιαστεί στον αφορά τι από 6,5 δι ευρώ ε, για 25 εκατομμύρια ανθρώπους πριν 10 χρόνια στα 24 δισεκατομμύρια να βοηθήσουμε 134 εκατομμύρια ανθρώπους φέτος. Αυτή είναι η αλλαγή των αναγκών. Θέλουμε να βάλουμε το στόχο 90 εκατομμύρια α, ανθρώπους στα προγράμματά μας το 2019. Δεν άλλαξαν οι βασικές συνιστώσεις των προσπαθειών. Αυξάνουμε τις προσπάθειες σε διάφορους τομείς Έχουμε βάλει προτεραιότητε όσον αφορά τι υποχρεώσει την προστασία των αμάχων, για την προστασία των εκτοπιστέντων και να ενισχυθεί θέση των γυναικών και των κοριτσιών μέσω διαφόρων πολιτικών και μέσω συμβουλών και προσανατολισμών. Άλλη προτεραιότητα. Να ξεπεράσουμε τη, δια, τη διαφοροποίηση μεταξύ ανθρωπιστικής βοήθειας και αναπτυξιακής βοήθειας και των διαφόρων φορέων. Και υποχρεώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας να βασίζονται να... μέσω άμεσης χρηματοδότησης των ντόπιων αρχών. Όπως είπε και ο κ. Στυλιανίδης, ακολουθήσουμε την προσέγγιση σε ντόπιο επίπεδο. Είναι αποτελεσματικότερο αυτό. Οι πιο καινοτόμε λύσεις προέρχονται από, τη... από τους τοπικούς φορείς. Δημιουργούμε και ντόπιο δυναμικό και έτσι έχουμε πιο εύκολη μετάβαση προς την ανάπτυξη. Και διάφοροι φορείς του ΟΗΕ θέλουν να συνεργαστούν περισσότερο τώρα πια έχουμε πιο κοινέ προσεγγίσεις, εντοπίζουμε καλύτερα τις ανάγκες, προγραμματίζουμε καλύτερα τις ανάγκες σε ρευστό, ομαδικά. Ο, ο Γενικός Γραμματέας Μάρκ Λάκοκ και η Ενιέτα Φόρ και ο Ντέιβιντ Μπίσλεϊ και είπατε, και είπατε, είπατε για τους πρόσφυγες θέλουν κοινό σύστημα για την κάλυψη των αναγκών. Θέλουμε να συναθρήσουμε την ανάλυση, την αξιολόγηση και τα δεδομένα μας ούτως ώστε να εφαρμόζουμε όλοι οι φορείς ε, με κοινό τρόπο τα προγράμματά μας. Αυξάνεται η συνεργασία. Περισσότερες ΜΚΟ θα συμμετάσχουν. Άρα θα αυξηθεί και η διαφάνεια όσον αφορά τη λειτουργία μας. Ενισχύουμε και τη δυνατότητα επαφής μας στην κοινωνία των πολιτών. Τι θέλουμε να κάνουμε, να βελτιώσουμε τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα. Η προσπάθεια ξεκίνησε το 2016. Πάνω από 60 κυβερνήσει, φορεί του ΟΗΕ και ΜΚΟ και η Διεθνή Συνομοσπονδία του Ερυθρού ε, Σταυρού και τη Ερυθρά Ημισελίνου και η Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού προσυπόγραψαν τη συμφωνία. Και αυτή η μεγάλη συμφωνία είναι ένα βήμα συζήτηση για αλλαγή. Από το 2016 έχουμε φέρει πολλέ βελτιώσει για τη χρηματοδότηση παρακολούθηση και συντονισμό ανθρωπιστική βοήθεια. Κάποια παραδείγματα. Αυτή η συμφωνία χρησιμοποιεί περισσότερο το ρευστό σαν ανταπόκριση, το είπε και ο Κ. Τηλιανίδη. Πολλέ μελέτε έδειξαν ότι είναι κάτι φθηνότερο, σε πολλέ περιπτώσει, φθηνότερο και πιο αποτελεσματικό. Από το 2015 τα προγράμματα σε ρευστό αυξήθηκαν κατά 40%. Φτάσαμε το 10% τη συνολική ανθρωπιστική βοήθεια Και κάποιοι ε, δωρητέ δίνουν περισσότερα χρήματα. Και τεχνολογία για τον ταυτοποίηση, βιομετρικά στοιχεία, μαζί με νέα μέσα καταγραφής συναλλαγών όπως το blockchain χρησιμοποιούνται στην Ιορδανία και την Τουρκία. Και έτσι οι πρόσφυγες μπορούν να καλύψουν τι ανάγκες τους και εμεί να μπορούμε να εντοπίσουμε την αποτελεσματικότητα τη βοήθεια καλύτερα. έχουμε αυξήσει ε, την ε, πολιτή ευέλικτη χρηματοδότηση. Όταν παρατείνεται η κρίση, ξεπερνάμε τον κύκλο το 12 μήνο. Κάποιοι δωρητές πήγαν από 15% σε 50% την πολιτική βοήθεια το 2017. Και άλλοι θα αυξήσουν τις εισφορές τους. Η συμφωνία μας μας οδήγησε να κάνουμε περισσότερα, να χρηματοδοτήσουμε άμεσα εθνικούς φορείς να δίνει τη βοήθεια σε τοπικό επίπεδο, στο του δυνατού. Μέχρι τώρα, από το συνολικό πόρου τη Ότσο, η εθνική ΜΚΟ, εθνικές ΜΚΟ, από το 6% που ήταν το 2015 αυξήθηκαν στο μερτικό των χρημάτων που παίρνουν αναχώρα. 204 εκατομμύρια δόθηκαν το 2017 σε εθνικές ΜΚΟ. Σύμφωνα με τις που αναλάβαμε, οι φορεί διάφοροι βελτιώνουν διατομιακέ ανάγκε και αξιολογήσει διατομιακών αναγκών για να λαμβάνονται στατικέ αποφάσει για συλλογική αντίδραση και χρηματοδότηση σε περίπτωση κρίση. Μετά την εκκίνηση του προγράμματο, κάναμε βήματα να προχωρήσουμε όσον αφορά τι δικέ μα υποχρεώσει. Τι εντάξαμε στη στρατηγική 2018-2021. Εσωτερικά προσπαθήσαμε οι υποχρεώσει αυτή τη συμφωνία να λαμβάνονται υπόψη στι διεργασίε μα και όχι στα σημεία ε, επαφή Θέλουμε να τους επιτόπιους φορείς να τους βοηθήσουμε. Βελτιώσουμε το δικαίωμα έφεσης να συμμετάσχουν οι ντόπιοι που πλήττονται από την κρίση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων περισσότερο. Αυτό θέλουμε. Βελτιώνοντας τις πρακτικές, ανοίγουμε το δρόμο για τις αναγκαίες αλλαγές και προσαρμογέ για το σύστημα τετροπιστική βοήθειας. Τρία χρόνια μετά την πρωτοβουλία που ξεκίνησε, πρέπει να δούμε πόσο οι διάφορα οι, θεσμικοί, οι θεσμοί μα έχουν πετύχει του στόχου που είχαμε θέσει. Πώ θα είναι βιώσιμη η προσπάθεια και ποια η κληρονομιά τη μεγάλη Συμφωνίας, επί τη οποίας βασιστήκαμε, τη μεγάλη συμφωνία. είναι η καλύτερη βάση για επίλυση προβλημάτων. Ναι, τα προβλήματα θα παραμείνουν. Ποτέ δεν θα έχουμε τέλειο σύστημα. Είναι εξαιρετικέ οι καταστάσει εργαζόμαστε και που παράγονται από τις κρίσεις, τις συγκρούσεις και τις φυσικές καταστροφές. Δεν υπάρχει άλλη πλατφόρμα ούτως ώστε να συναθρίζονται όλοι οι φορείς και να βγαίνουν στη σκηνή μαζί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν μεγάλο δωρητή, θα πρέπει να εφαρμόσει αυτή τη μεγάλη συμφωνία και τη σχετική πρωτοβουλία για να αντιμετωπίσουμε τα εμπόδια, για να εφαρμόσουμε πλήρως τη συμφωνία και να χρησιμοποιήσουμε το δυναμικό που περιέχει να υπάρχει καλύτερη, ε, καλύτερος του κινδύνου μεταξύ των φορέων και των δωρητών. Πολύ δίνουμε στους εθνικούς εταίρους τους κινδύνους, στις εθνικές ΜΚΟ που είναι στην πρώτη γραμμή και αντιμετωπίζουν ως κινδύνους. Πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ δωρητών και των εφαρμοστικών φορέων και το δικαιωτικό άχθος να μειωθεί για να είμαστε πιο αποδοτικοί. Μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μέσω συλλογικής δράσης και μόνο με συμμετοχή και των μελών του Ευρωκοινοβουλίου. Επιτρέψτε μου να πω λίγα λόγια. Για αυτά που είπε ο αναπληρωτής γραμματέας Μάρκ Λέκοξ για τη βελτίωση του συστήματος. Αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των εμπλεκομένων μερών στη σύραξη. Γιατί αυτοί οδηγούν στην αναγκαστική μετακίνηση πληθυσμών. Καλύτερο σύστημα χρηματοδότησης, καλύτερο συντονισμός να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε υψηλέ προδιαγραφέ επαγγελματισμού που ακολουθούμε στι δράσει μα. Να αυξήσουμε τι προσπάθειε για να επηρεάσουμε τη συμπεριφορά των εμπλεκομένων, να εφαρμόζονται καλύτερε πρακτικέ εκεί που υπάρχουν συγκρούσεις του τελευταίους μήνες. Προσπαθούμε να συντονίσουμε καλύτερα τις συνιστώσεις για να ε, έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Θέλουμε καλύτερους επαγγελματίες επιτόπου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Πώς ανταποκρινόμαστε μετά οικονομικά στα προβλήματα. Τώρα είμαστε αντιδραστικοί, αντιδρούμε. Καλύτερο σύστημα θα ήταν να έχουμε διαπραγματεύσει εκ των προτέρων να έχουμε συμφωνήσει πριν και μετά, να, άμα συμβεί κρίση, να δίνουν τα χρήματα κατευθείαν που έχουν προσημειωθεί και να αντιμετωπίζουμε και θέματα όπως η ξηρασία. Μικρά νησιά ε, προσπαθούν να αντιμετωπίσουν μεγάλες φυσικές καταστροφές και τα έκτακτα προϊόντα που δίνουν οι αναπτυξιακές τράπεζε όλο και σε περισσότερου δανειστές για αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Έτσι θα σωθούν περισσότερες ζωές, θα μειώσουμε τις ανθρωπιστικές κρίσεις και ίσως εξαλείψουμε τι ανθρωπιστικέ κρίσει. Θα μειωθεί το κόστος και θα υποστηρίξουμε αποτελεσματικότερα καλύτερε προσπάθειες. Με πολλοί φορεί του ΟΗΕ, αρχίζουν να εθετούν αυτές τις προσεγγίσεις εκ των προτέρων κανονισμένες. Πέρα συνεργασία στην ανθρωπιστική βοήθεια, όπως είπε ο κ. Στυλιανίδης, συνεργαζόμαστε με την Παγκόσμια Τράπεζα, με την ΕΚΟ, με το UNDP, για να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε κοινέ αξιολογήσεις αναγκών και κοινή ανάλυση. Και ελπίζουμε ότι τελικά αυτό θα γίνει κανονικός τρόπος λειτουργίας παντού. Θα βρείτε μέρη όπου οι αναπτυξιακοί φορεί παίζουν μεγαλύτερο ρόλο για την μείωση των προβλημάτων. Επέστρεψα από το Μαλί. Υπάρχει πιθανότητα ότι με τη διασύνδεση ανθρωπιστική βοήθεια και νευτική διαδικασία να αποφύγουν μεγαλύτερε κρίσει πολλέ από τι επιτροπέ στο Μαλί, κυρίω στις περιοχέ που αντιμετωπίζουν ξηρασία, αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα. Όπω ήταν η κρίση του 2003, με σωστή υποστήριξη αναπτυξιακή βοήθεια, όχι μόνο ανθρωπιστική βοήθεια και με διάλογο και ειρηνευτική διαδικασία μπορούμε να αποφύγουμε παρόμοιε κρίσει να ξεσπάσουν στο Μαλί ε, όπω παλιά και στη γενικότερη, στην ευρύτερη περιοχή. Θέλουμε να βελτιώσουμε το σύστημά μα, τι δομέ μα για να αποφευχεί η σεξουαλική εκμετάλλευση και η κακομεταχείριση. Είδαμε πολλέ εκθέσει από τέτοια συμβάντα και καταγγελίε, και είναι καθημερινό φαινόμενο για πολλού ευάλωτου πληθυσμού υπό την ηγεσία της Ενριέτα Φιόρ που είναι εκτελεστικό μέλος της UNICEF βελτιώνουμε τους μηχανισμούς καταγγελιών για να κινούμεθα έγκαιρα και να κινούμεθα κατά εκείνων που βιοπραγούν. Επέστεψα από την εμπειρία που είχα σαν συντονιστής για την κρίση στη Συρία στον Καζιατέπ και πολλές από τις συμφωνίες που έχουμε κάνει λειτουργούν επί τόπου. Η ντόπια αντιμετώπιση έχει μεγάλο αντικτύπο. Οι Συριακές ΜΚΟ είναι πολύ αποτελεσματικότερες στο να βοηθούν τον πληθυσμό και τις κοινότητες και είναι καινοτόμες στον προγραμματισμό. Έχουμε υπέροχη ευκαιρία μέσω τοπικών φορέων να κινηθούμε, να τους ενισχύσουμε, το τοπικό δυναμικό να βελτιωθεί και να γίνουν βιώσιμα τα προγράμματα. Η ηγεσία τους στο συντονισμό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα. Πρέπει να βασιστούμε επί αυτών των μοντέλων και να προσανατολιστούμε βάσει αυτών, εκτός να κινούμεθα μόνο θεωρητικά σε επίπεδο αρχηγείου και να μην λαμβάνει υπόψη τις ντόπιε ανάγκες. Θα πάρουν παραδείγματα από το τοπικό επίπεδο και να προσανατολιζόμεθα. Ευχαριστώ για το χρόνο που μας δώσατε και για την τεράστια υποστήριξη που δώσατε στις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ. Thank you, Και τώρα περνάμε σε παρεμβάσεις από εκπροσώπους κοινωνίας των πολιτών. Είμαι Βάσκεφ πρώτα απ' όλα, εκπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή, Επιτρο... στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ των ε, γιατρών χωρίς σύνομα. σύνορα. Ευχαριστώ που μας παρακαλέσατε. Entertainment here because ε, we don't share all the aspects or all the views that have been ε, Άκουσα τι πολύ καλέ προτάσεις που παρουσιάσαν. Θα ήθελα να κάνω μια γενική παρουσίαση. Δύο προκλήσεων που νομίζουμε ότι είναι πολύ σημαντικέ σήμερα στους γιατρού χωρίς σύνορα και να απαντήσω σε κάποια σχόλια που έγιναν και να εξηγήσω κάποιες από τις απόψεις μου που είναι κάπως διαφορετικές. Και επίσης γιατί δεν είμαστε τι βγαίνει στα πλαίσια της διάσκεψης κορυφής. Όσον αφορά τις προκλήσεις σήμερα, το σημείο κινησής μας είναι, είναι ότι στην πράξη το δίκαιο που διέπει την ε, ανθρωπιστική βοήθεια δεν είναι του επίπεδου που θα πρέπει. Πιστεύουμε λοιπόν ότι Περισσότερο από ποτέ θα πρέπει κάτι να κάνουμε. Επιτόπου όμως βλέπουμε ότι η ισχύουσα νομοθεσία δεν γίνεται σεβαστή και δεν υπάρχει πολιτική βούληση, δέσμευση να γίνουν αλλαγές. Για να γίνουν αλλαγές θα πρέπει να υπάρχει αξιοπιστία. Αξιοπιστία τι σημαίνει, θα πρέπει να γίνουν ανεξάρτητες έρευνες και με τα μέσα που προσφέρει η Σύμβαση της Γενέβης. Πράγμα που δεν συμβαίνει, επαναλαμβάνω. Θα μιλήσω για δύο θέματα που εμείς καλούμε εγκληματικο... Um, uh, ποινικοποίηση της ανθρωπιστικής ε, ε των, του τι ακριβώς συμβαίνει πολλές φορές στα πλαίσια της χορήγησης της ανθρωπιστικής βοήθειας. Δεν θα αναφερθώ στις διάφορες επιθέσεις που έχουν γίνει, αλλά στα επιχειρήματα που χρησιμοποιούν για τη δικαιολογήσουν. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα επιχειρήματα αυτά έχουν σχέση με την ε, αφήγηση, νομοθεσία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Στο Αφγανιστάν, όταν στο Κοντούς έγινε επίθεση ειδικών δυνάμεων στο νοσοκομείο, όλα ελέγχθη ότι έγιναν στα πλαίσια της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Οι δυνάμεις αυτές χρησιμοποίησαν το δικό του τρόπο και όλη η πόλη του Κουντούς με 900.000 πολίτες πληθυσμό θεωρήθηκε εχθρικό έδαφος. So there was not, for example, there was no uh, assessment of the proportionality. λοιπόν για την επίθεση ε, χωρίς καμία των προτέρων προειδοποίηση ειδικές δυνάμεις στα πλαίσια της ε, επίθεσης κατά της τρομοκρατίας. Επίσης, στην Ιεμένη πρέπει να πω ότι έγιναν επιθέσεις σε πέντε εγκαταστάσεις των ε, γιατρών χωρίς Και στις τέσσερις περιπτώσεις δικαιολογείται αυτή η επίθεση από ό,τι πρέπει να πω ότι σε μία περίπτωση έμπαινε ένα αυτοκίνητο στο νοσοκομείο, εξεράγει μία βόμβα, εννέα θανάτους είχαμε, πέντε παιδιά, ένα γιατρό και η δικαιολογία ήταν ότι υπήρχε κάποιος στόχος ο οποίος έπρεπε να καταστραφεί μέσα στο αυτοκίνητο. Δυσανάλογα όλα αυτά και καμία σχέση δεν έχουν με την ε, ανθρωπιστική βοήθεια. Και θεωρήθηκε η καταστροφή μεγάλους μέρους αυτού του νοσοκομείου ως ε, underground Παρά ως παράβρευρη απώλεια. Fight against Στην Ιγυρία. Δεν θα δώσω περισσότερα παραδείγματα από αυτό. το 2017 βομβαρδίστηκε ένα καταβλισμός, 19 νεκρούς είχαμε, με επιχείρημα ότι υπήρχε ε, απειλή επίθεσης εκ μέρους της Μπόκο Χαράμ. Τι σημαίνουν όλα αυτά. Ότι αυτά που συμβαίνουν, αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι ότι σε περίπτωση που έχουμε μία κατάσταση σύγκρουσης και διένεξης και σε περιοχές που δεν υπάρχει έλεγχος σοβαρός, δεν υπάρχει πρόσβαση σε νοσηλεία, σε νοσοκομεία για τον απλό κόσμο. Δεν υπάρχει πρόσβαση, αν υπάρχει είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Επίσης, κάτι το οποίο είναι ενισχυτικό είναι το εξής. Η ιατρική βοήθεια που παρέχεται από τους γιατρούς χωρίς σύνορα θεωρείται από πολλούς ηλική υποστήριξη προς τους ε, τρομοκράτες. και κυρίως βρίσκονται σε μεγάλη πίεση οι, τα άτομα που προέρχονται από τη χώρα στην οποία δραστηριοποιούμαστε για συνεργασία. Πιστεύω λοιπόν ότι στα πλαίσια αυτού που αναφέρθηκε και προηγουμένως για τον Nexus Dynamics θα πρέπει να κάνουμε κάτι περισσότερο ώστε να μπορέσουμε στα πλαίσια των δραστηριοτήτων μας και της, ε, της ε, ανθρωπιστικής βοήθειας και αρρωγής να είμαστε πιο ενωμένοι και με πάρα πολύ ε, αποτελεσματικό τρόπο να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία. Δεν ξέρω αν σας τα εξηγώ αυτά σωστά. Η ποινικοποίηση της ε, βοήθειας στα πλαίσια των προσφύγων και μεταναστών. Θα αναφέρω το παράδειγμα του Ναουρού, μιας μικρής νησίδας στην Οκεανία. Δουλέψαμε εκεί για 11 μήνες για να βοηθήσουμε σε θέματα ψυχικής υγείας και πέρσι το φθινόπωρο μας ζητήθηκε να αποχωρήσουμε μέσα σε 24 ώρες έπρεπε να φύγουμε. Είχαμε 124 ασθενείς με τάσεις αυτοκτονίες και κάποιους που έπρεπε να πάρουν ψυχιατρική βοήθεια. Κατορθώσαμε κάποιους να σχέση που τους βοηθάνε μέσω της τηλεϊατρικής, αλλά το περασμένο Σαββατοκύριακο μάθαμε ότι απαγορεύτηκε και αυτό στο Ενούρου. Άρα δεν μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Επίσης, υπάρχει μία επιστολή στην οποία σχολιάζεται η παρουσία μας εκεί. Επίσης, τα πλαίσια της έρευνας και διάσωσης στην ε, Μεθόγειο, Μεσόγειο. Για μας πρόκειται για δραστηριότητα διάσωσης ανθρωπίνων ζώων είναι κάτι το οποίο αφορά ανθρωπιστική βοήθεια, βοήθεια προς ανθρώπους, αλλά σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες μας κατηγορούν κάποιοι για παράνομη διακίνηση αποβλήτων στα πλαίσια της Και για μας πρόκειται για προσπάθεια να σταματήσει η παροχή ανθρωπιστικής ενίσχυσης και βοήθειας που παρέχομαι. Διότι αυτό που... πρόκειται για κάτι το οποίο λαμβάνει πολιτική διάσταση αυτό που κάνουμε και για μας αυτό είναι πρόβλημα είναι έλλειψη αναγνώρισης της ανεξαρτησίας της ανθρωπιστικής δράσης και όλων των δραστηριοτήτων διάσωσης ζώων. Στην αρχή εξηγούσα ότι η MSF απεφάσισε στο τέλος, δεδομένου ότι συμμετείχαμε στην ε, διαδικασία να μην συμμετάσχουμε στην σχετική διάσκεψη κορυφής, δύο ήταν τα επιχειρήματά μας. Πρώτα απ' όλα, ο περιεχόμενο των θεμάτων προς ελαχιστοποιούσε την ε, ευθύνη του κάθε κράτους και η, για μας η έννοια, η αντίληψη της ανθρωπιστικής βοήθειας δεν ήταν η ίδια με την δική μας. Πρόκειται για κάτι το ιδιάζον, πρέπει να το σεβόμαστε και θα σας το εξηγήσω με ένα παράδειγμα. Πρέπει να τελειώνω δυστυχώς. Η ανταπόκριση στην έμπολα. Πρόκειται για ένα πρότυπο αντίδρασης σε κάθε τοπικό επίπεδο συγκεκριμένα και με κάθε Υπουργείο Υγείας και συντονισμένα με τους εκπροσώπους της ανθρωπιστικής βοήθειας. Αλλά πολλές φορές, για να δώσω ένα παράδειγμα, στο Κίμπου δεν γίνεται τίποτα αποτελεσματικό, δεδομένου ότι είμαστε σε μία ζώνη σύγκρουσης και πολλοί εξέφρασαν την δυσπιστία τους, δεδομένου ότι όλη η καμπάνια γίνεται υπό την αιγίδα της κεντρικής κυβέρνησης Αλλά πιστεύουμε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δημιουργεί δυσπιστία για τον τρόπο με τον οποίο συντονίζονται τα πράγματα και είναι κάτι που θα μας φέρει πολύ περισσότερα κρούματα, κρούσματα. Λυπούμε, αλλά πρέπει να πω ότι πολλές φορές η ανθρωπιστική αξία δεν μπορεί να έχει, για να χρησιμοποιήσει ένα οικονομικό όρο, αυτή την σχέση κόστους-οφέλους που χρησιμοποιείται. Επίσης, για την ε, για το παράδειγμα της, ε, της Κεντρικής Αφρικής. Χρειάστηκε σε μια συγκεκριμένη περίπτωση να στείλουμε ένα τσάρτερ για να παρέχουμε βοήθεια, το οποίο ήταν κάτι το πολύ δαπανηρό για να αντιμετωπιστούν επίγουσες ανάγκες, χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον τρόπο μεταφοράς. Άρα πρέπει και να είμαστε πολλές φορές προσεκτικοί με το θέμα του κόστους απόδοσης. Αλλά να λάβουμε υπόψη το γεγονό ότι η ανθρωπιστική δράση λαμβάνει χώρο σε δύσβατες περιοχές, σε δύσκολες συνθήκες και επίσης να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι είναι κάτι το πολύ επικίνδυνο και δαπανηρκρό να στείλει κάποια εταιρεία ένα τσάρτερ εκεί. Τώρα, όσον αφορά το cash. Καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι. Αλλά είναι σημαντικό όταν αναλαμβάνετε του είδους δραστηριότητες να είστε θέση να ελέγχετε το ότι ο, τα άτομα τα οποία πρέπει να λάβουν αυτό το cash έχουν πρόσβαση σε αυτή την υπηρεσία που παρέχεται. Έχουμε παραδείγματα στα οποία οι πρόσφυγες είναι θύματα διάκριση όταν πηγαίνουν στους, ε, στα δημόσια ιατρία, ακόμη και όταν έχουν μαζί τους αυτές τις κάρτες cash. Θα σταματήσω εδώ. Gracias. Πολύ. Τώρα θα δώσουμε το λόγο σε εκπροσώπους της ίδιας οικογένειας, ο καθένας όμως τον κλάδο του. Πρώτα απ' όλα, στην, ε, ε, στον εκπρόσωπο του Ερυθρού Σταυρού και εκπρόσωπο του Ερυθράς Ημισελίνου. Δεν χρειάζεται να καθυστερήσω περαιτέρω για να πω πόσα οφείλει η ανθρωπιστική βοήθεια στον Ερυθρό Σταυρό από ιστορικής πλευράς και σήμερα, τη στιγμή κατά την οποία ε, ορτάζουμε και την 70η επέτειο της Σύμβασης της Γενέβης. Ο κύριος Φούλτεμαν πρώτα απ' όλα θα λάβει το λόγο που είναι από το 2015 στο Βέλγιο μέλος του Ερυθρού Σταυρού και έχει πείρα σε πάρα πολλές χώρες, στην Κροατία, στην Καράγουα, σε πόρες της Αφρικής και βεβαίως στη Νέα Υόρκη, στα γραφεία του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού. Ευχαριστώ πολύ, Δον Ενρίκε. Ε, Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Αγαπητοί Πρόεδρε, αγαπητοί Ευρωβουλευτές, μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης, αγαπητοί συνάδελφοι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σας ευχαριστώ που μας προσκαλέσατε σε αυτή την τελευταία δημόσια ακρόαση και προτού ξεκινήσουν τα 8 μου λεπτά θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω εκ μέρους του ICRC όλους σας για τη διπλωματική και οικονομική βοήθεια και στήριξη που μας παρέσχε η Ευρωπαϊκή Ένωση στη διάρκεια της τελευταίας θητείας. Και μας ενθαρρύνει πάρα πολύ το γεγονός ότι ακούσαμε ότι σκοπεύετε να αυξήσετε μάλιστα τα κονδύλια για την ανθρωπιστική βοήθεια στο επόμενο ΠΔΠ. Θέλω να επικεντρωθώ σε τρεις τομείς που άπτονται της ανθρωπιστικής βοήθειας στο μέλλον και θα διανύμουμε και στους ευρωβουλευτές ε, ηλεκτρονικά αντίτυπα της δικής μας στρατηγικής του ICRC για την περίοδο 2019-2022 που έχουμε αναπτύξει και που πιστεύω ότι μπορεί να συμβάλλει και στη συζήτηση που γίνεται εδώ. Σίγουρα εμάς μας βοηθά στο να ε, διαμορφώσουμε τον δικό μας ε, προσανατολισμό. Θεωρώ ότι μπορεί να υπάρξει σύγκληση μεταξύ ICC και Ευρωπαϊκής Ένωσης στις δράσεις τους τα επόμενα χρόνια. Να ξεκινήσω με ορισμένα ε, αριθμητικά στοιχεία. Γίνεται πολύ συχνά λόγος ε, για τις συγκρούσεις και φυσικά εκεί κατευθύνεται η ανθρωπιστική βοήθεια κατά κύριο λόγο. Οι 20 μεγαλύτερες ανθρωπιστικές κρίσεις αυτή τη στιγμή στον κόσμο ε, αντιστοιχούν στο 80% των ε, ε, αναγκών ανθρωπιστικής βοήθειας που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Καταλαβαίνετε δηλαδή την κλίμακα αυτών των κρίσεων και τις ανάγκες που δημιουργούν αυτές οι κρίσεις. Και πιστεύουμε ότι οι συγκρούσεις αυτές θα συνεχίσουν τα επόμενα χρόνια να μας απασχολούν. Από αυτή την άποψη λοιπόν η παγκόσμια στάθεια, η ευθραυστότητα ο εκτοπισμός αλλά και τα μακροχρόνια προβλήματα που προκαλούνται στις κοινωνίες και στα κοινωνικά συστήματα είναι κάτι που πρέπει να ειδωθεί και από την ανθρωπιστική και από την αναπτυξιακή και φυσικά και από την πολιτική σκοπιά. Ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι υπάρχει τάση που δείχνει ότι το χάσμα ανάμεσα στις ανάγκες και στη βοήθεια που δίνεται μεγαλώνει. Όταν προετοιμαζόμουν για τη σημερινή εκδήλωση, διάβαζα και διάβασα κάπου ότι ο συνολικός ε, προϋπολογισμός ανθρωπιστικής βοήθειας ανέρχεται σε περίπου 30 δισεκατομμύρια, που είναι ποσό ίσο με αυτά που ξοδεύει ο κόσμος, ο πλανήτης, σε τσίχλες κατέτος. Οπότε ίσως αυτό σας δίνει ένα στοιχείο για το πόσα τελικά δίνονται. Ανέφερε ο Ενρίκε ότι σήμερα συμπληρώνονται, φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια από την υπογραφή της διακήρυξης της Γενέβης για τα δικαιώματα των προσφύγων. Και θα συμφωνήσω και εγώ ότι σε πάρα πολλά τμήματα του κόσμου υπάρχει παραγνώριση ε, της ανάγκης ε, για ανθρωπιστική βοήθεια που είναι και αιτία αλλά και σύμπτωμα της βίας. Αυτή είναι η αρνητική πλευρά. Υπάρχει όμως και μια θετική πλευρά της νομοθεσίας για την ανθρωπιστική βοήθεια της γενέβη. Και αυτό είναι το ότι μπορούμε πραγματικά να, να ισχυριστούμε ότι έχουν σωθεί εκατομμύρια ζωή, ζωές, έχουν μετριαστεί αρνητικές επιπτώσεις για εκατομμύρια ανθρώπους. Αυτό που μπορεί λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κάνει είναι να, να ξαναδηλώσει την ε, προσήλωσή του στην προστασία των αμάχων, την ε, την ανθρώπινη μεταχείριση των κρατουμένων και των ομήρων. Υπάρχουν δε κάποια προβλήματα τα οποία επιτείνονται ακόμη περισσότερο, υπερ, υπερπληθισμός, αστικοποίηση, κλιματική αλλαγή, άνηση οικονομική ανάπτυξη. Το ζητούμενο εδώ και το, το, το, η ουσία μάλλον του θέματος είναι ότι κανένας τομέας μόνος του δεν μπορεί να απαντήσει στο βάθος και στο εύρος αυτών των ε, ανθρωπιστικών κρίσεων που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Αν θέλουμε λοιπόν να σημειώσουμε πρόοδο, χρειάζεται ισχυρή στήριξη όχι μόνο από εκείνους που, που ασχολούνται με τον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας αλλά και από κυβερνήσεις, από διεθνείς οργανισμούς και από την κοινωνία των πολιτών. Από τη δική μας πλευρά θα προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε εκείνο, το ανθρωπιστικό, εκείνο τον ανθρωπιστικό χώρο ώστε να μπορεί να παρέχεται βοήθεια αλλά και, και επιμένω σε αυτό, την προστασία των πολιτών που έχουν πληγεί από ε, συγκρούσεις. Όσον αφορά τη σύγκληση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ημών, με ΙΤΑ, αυτή υπάρχει σε τρεις τομείς. Στην ομοθεσία για την ανθρωπιστική βοήθεια, τη βιωστημότητα των αποτελεσμάτων που επιτυχάνονται και τέλος, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό που αποκαλούμε ψηφιακή μετάβαση για, την πρώτη, για τον πρώτο τομέα που ανέφερα, την ομοθεσία, το δίκαιο. Πρέπει να συνδέσουμε ξανά το δίκαιο με τις αρχές μας. Το ανθρωπιστικό δίκαιο περιλαμβάνει εχέγγυα για να εξασφαλίζεται η αμερόλεπτη ανθρωπιστική δράση. Και από αυτή την άποψη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συντάξει τις δικές της κατευθυντήριες γραμμές για την ε, συμμόρφωσή της με το Διεθνές Δίκαιο για την Ανθρωπιστική Βοήθεια. Έχει δηλαδή με άλλα λόγια χαράξει ένα δικό της πλαίσιο ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται και να συμμορφώνεται με καλύτερο τρόπο στο Διεθνές Δίκαιο για την Ανθρωπιστική Βοήθεια. Θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό έγγραφο, ένα πολύ σημαντικό εργαλείο αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές γιατί βλέπουμε ότι πολλά κράτη-μέλη ε, έχουν υποστηρίζουν πλέον περισσότερο κρατικούς και μη κρατικούς φορείς κατά την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί ε, πρέπει να σημειώσουμε ότι ο σεβασμός στο, στο δίκαιο είναι πάρα πολύ σημαντικός. Επίσης θέλω να εξάρω την οδηγία του 2017 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας όπου αναφέρεται ρητός ότι πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή της ποινικοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Πρέπει λοιπόν με ανησυχία να σας ε, ενημερώσω ότι πολλές φορές περιορίζεται η ανθρωπιστική βοήθεια με το πρόσχημα αντι, της αντιτρομοκρατίας ή άλλων κυρώσεων, ενώ στην πραγματικότητα ο, ο αντίκτυπος αυτών των μέτρων ε, τελικά ε, πλήττει κυρίως τις ανθρωπιστικές οργανώσεις, τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ελπιδρούν. και να παρέχουν την βοήθεια. Και έτσι πλήτεται, πλήττονται και εκείνοι που παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια και εκείνοι στους οποίους απευθύνεται, για τους οποίους προορίζεται η ανθρωπιστική βοήθεια. Από αυτή την άποψη, εμείς πιστεύουμε ότι είναι εφικτό να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ της απολύτως δίκαιης και βάσιμης ανάγκης των κρατών να καταπολεμήσουν την ε, τρομοκρατία να προλάβουν τρομοκρατικές επιθέσεις. Είναι βεβαίως απολύτως θεμητό αυτό από την πλευρά των κρατών, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνεται ε, με ταυτόχρονη τήρηση των αρχών που διέπουν την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Επίσης θέλω να τονίσω σήμερα το απόγευμα εδώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την την, έχει καταλήξει σε συνένεση όσον αφορά την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το υπενθυμίζουμε αυτό. Ε, η ευρωπαϊκή αυτή συνένεση περιλαμβάνει ξεκάθαρη δέσμευση ε, και προσήλωση στις ανθρωπιστικές αρχές και ορίζει επίσης ότι η ανθρωπιστική βοήθεια δεν μπορεί από μόνη της και καθεαυτήν να γίνει εργαλείο για την ε, καταπολέμηση των ανθρωπιστικών κρίσεων. Και αυτό συνδέεται και με το τρίπτυχο που αναφέραμε. Τέταρτος τομέας, βιώσιμη ανθρωπιστική βοήθεια και αντίκτυπος. Είναι ζωτική σημασία αυτή η πτυχή. Είναι ζωτική σημασία και για τη δική μας στρατηγική, γιατί βλέπουμε ότι οι έκτακτες ανάγκες αυξάνονται από τις κρίσεις δηλαδή. Ταυτόχρονα όμως έχουμε να αντιμετωπίσουμε μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των κρίσεων στην αξιοπρέπεια, την προστασία, την ασφάλεια των πληθυσμών. Οι προκλήσεις λοιπόν που αντιμετωπίζουμε τόσο ως, ανθρω... ως ανθρωπιστικές οργανώσεις αλλά και ως ε, ε, ευρωπαϊκοί θεσμοί εσείς είναι αυτό το παραδοσιακό ανθρωπιστικό μοντέλο, το παραδοσιακό χρηματοδοτικό μοντέλο δεν είναι προσαρμοσμένο δεν είναι προσαρμοσμένα σε αυτήν την ε, βιώσιμη διάσταση, σε αυτήν την βιώσιμη προσέγγιση. Στην πραγματικότητα είναι προσελωμένο πάντοτε στο μοντέλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα δικά μας στο να δίνονται απαντήσεις άμεσες όταν ξεσπούν κρίσεις. Αντιθέτως λοιπόν εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να βρεθούν τρόποι ώστε να εξασφαλίζονται και βραχυπρόθεσμες ε, ε βοήθεια, αλλά να εξασφαλίζεται και ε, να εξασφαλίζεται και η χρηματοδότηση μακροπρόθεσμων στρατηγικών και μέτρων, όπως για παράδειγμα στην εκπαίδευση, όπως είπε ο Επίτροπος στη, στη Λιανίδης. Και αυτό θα πρέπει να είναι μια διάσταση που θα πρέπει να την υπόψη από τον σχεδιασμό κιόλας των προγραμμάτων και φυσικά και στην υλοποίηση. Υπάρχει λοιπόν μια σαφής διασύνδεση μεταξύ βραχυπρόθεσμων αναγκών και μακροπρόθεσμων επενδύσεων. Γι' αυτό και καλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση με ευέλικτο και πολιετή προγραμματισμό να εντάξει και αυτή τη διάσταση στον δικό της, στη δική της πολιτική και ε, να σας ενημερώσω με αυτή την ευκαιρία ότι εμείς ήδη έχουμε ξεκινήσει ε, έναν αντίστοιχο πολιετή προγραμματισμό για διάφορες χώρες της Μέσης Ανατολής. Τέλος, θέλω να αναφερθώ στην ψηφιακή μετάβαση, για την οποία ε, έχουν υποθεί πολλά. Πολλά υπόθηκαν σήμερα επίσης και για, το ρευστό, για τα μετρητά ε, και το πόσο σημαντικό εργαλείο είναι. αλλά θέλω να σταθώ και στο πόσο σημαντικό εκεί είναι η ψηφιακή μου βοήθεια, η μετάβαση, πόσο έχουν βοηθήσει τι ανθρωπιστικές οργανώσει, και θα πρέπει το, το ίδιο η ψηφιακή αυτή μετάβαση να αφορές, να ε, καλύψει και, ε, και τα μετρητά που δίνονται ως βοήθεια στους ε, πληγέντες ανθρωπιστικών κρίσεων. Στο πλαίσιο αυτό, εμείς έχουμε ε, συντάξει και ένα ε, εγχειρίδιο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της ψηφιοποίησης. Γιατί όσο πιο πολύ ψηφιοποιούνται τα πράγματα, τόσο αυξάνονται και συγκεκριμένοι κίνδυνοι. Εμείς λοιπόν ε, συντάξαμε ένα σχετικό εγχειρίδιο για να βρεθήσουμε τι ανθρωπιστικέ οργανώσει στην ε, διαδικασία αυτή τη ψηφιακή μετάβαση. Τέλο, υπάρχει ενωσιακή στρατηγική για την ανθεκτικότητα και την προηγούμενη εβδομάδα εγκρίθηκαν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την κλιματική διπλωματία. Είναι και αυτά πολύ σημαντικά έγγραφα για τι μελλοντικέ μα εργασίε. είναι διευθυντής ε, του Γραφείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Ερυθρού Σταυρού και της ε, Διεθνούς Ομοσπονδίας Ερυθρού Σταυρού και ε, της ε, Ερυθράς Ημισελίνου. Ντονί, έχει το λόγο. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Γκερέρο. μεγάλη χαρά για μένα να έρθω εδώ και σας μιλήσω για την άποψη του Ερυθρού Σταυρού για το μέλλον τη ανθρωπιστική βοήθεια. Θα εστιαστώ επί δύο πτυχών. Αυτέ αναφέρθηκαν από προλαλήσαντε. Η ντόπια αντιμετώπιση, η επιτόπια αντιμετώπιση και μετά ο συσχετισμο με την αναπτυξιακή βοήθεια. Πολύ σημαντικό για τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται καθημερινά ο Ερυθρό Σταυρό και οι φορεί του Ερυθρού Σταυρού. Παράδειγμα, το Μπαγκλαντέ. Η Ερυθρά Έλληνο του Μπαγκλαντέ επί σειρά ετών δίνει ιατρικές υπηρεσίες σε ευάλωτες κοινωνίες, συνεργάζεται και με θελοντές των κοινοτήτων προς βελτίωση της ετοιμότητάς τους για κυκλώνες και πλημμύρες. Το Μπαγκλαντέσα χώρα ε, είναι πολύ επιρρεπές σε φυσικές καταστροφές και επί 18 μήνες φιλοξενεί εκτοπιστέντες υπηκούς του Μιανμάρ, πάρα πολλούς με την υποστήριξη αρχικών εθνικών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Στο Κόξ Μπαζάρ έχετε έρθει κάποιες αποστολής στον Μπαγκαντέ και ο Φιλανδικό Ερθοσταυρό και ο Γερμανικό Ερθοσταυρό, χάρη στη βοήθεια τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, έχει κινητά νοσοκομεία εκεί. Μπόρεσαν να αυξήσουν οι εθνικοί φορεί την ανταπόκρισή του και να επεκτείνουν τι δραστηριότητε του σε προγράμματα για βραχυπρόθεσμη χορήγηση ρευστού ιατρική βοήθεια για να βοηθήσουν εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπιστέντων που έχουν καταβλισμού στα σύνορα. Όσον αφορά την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και την αύξηση αντοχής των κοινοτήτων είναι στο επίκεντρο των προσπαθειών που καταβάλουν ο Ιθός Σταυρός και η Ερυθράη Η Ερυθράη Μισέλινος στον Μπαγκλαντές δίνει παραδείγματα και δείχνει το βασικό στόχο να αντιμετωπίζονται επιτόπου προβλήματα, να υπάρχει ανταπόκριση επιτόπια που θα είναι επιτόπια στο βαθμό του δυνατού, αλλά θα συμπληρώνεται από διεθνή ανταπόκριση στο βαθμό της αν... του αναγκαίου. Οι τοπικοί φορείς, και εδώ μιλάμε για τον Ερυθρό Σταυρό και τους εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, είναι εκεί πριν ξεσπάσει η καταστροφή, ετοιμάζουν τι κοινότητε να προετοιμαστούν κατά τη διάρκεια τη κρίση, παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια και πολλοί μετά αφού φύγουν οι διεθνείς φορείς συνοδεύοντας τις κοινότητες στην οδό προς ανάκαμψη. Συμφωνώ μαζί σας ότι αυτό θολώνει τις γραμμές μεταξύ του τι αποτελεί καθαρά βοήθεια για έκτακτη ανάγκη και μακροπρόθεσμη ε, αναπτυξιακή βοήθεια. Το Δεκέμβριο του 2018 ο Διεθνή Ερυθρό Σταυρό, εθνικέ εταιρείε, η Ερυφθά Έλληνο, ξεκίνησαν, ε, ετοίμασαν ένα έγγραφο κοινή θέσεω με συστάσει προ την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη σχετικά με τη συσχετισμό ανθρωπιστική βοήθεια και αναπτυξική βοήθεια. Και με μεγάλη απογοήτευση δική σα, δεν θα σα διαβάσω πλήρω το κείμενο, αλλά θα αναφέρω δύο-τρία σημεία που περιέχει το κείμενο που θεωρώ ότι είναι σημαντικά. Ο Ερυθρό Σταυρό τονίζει την ανάγκη ενισχύσεω τη σχέση μεταξύ ανθρωπιστικής και αναπτυξιακή συνεργασίας. Αυτό είναι ο κόμβο, αν θέλετε, τη διασύνδεση και το μοίρασμα πληροφοριών με αυτούς που ασχολούνται με νευτικές διαδικασίες σε περίπλοκες διεργασίες είναι δημιουργεί αποκατάσταση εμπιστοσύνη. Αυτό είναι ο τριπλός δεσμό χωρί να υπονομεύεται ανθρωπιστική αξία και να διευκολύνει την πρόσβαση στους πληγέντε πληθυσμού. Στην περίπτωσή μα καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό ισχύει και για άλλους εταίρου βεβαίως και άλλου δωρητέ, αλλά τώρα είμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μιλάμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, να παράσχει χώρο ευελιξία μπορείτε να το πείτε στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ενώσης και στα μέσα χρηματοδότησης για μη κρατικούς φορείς και κοινωνίες των πολιτών για να παίξουν το ρόλο τους ανταποκρινούμενοι στις ανάγκες αναπτυξιακής βοήθειας και ανθρωπιστικής βοήθειας και να κάνουν το συσχετισμό μεταξύ ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής δράσης. Κάτι απαραίτητο. Φέτος, όπως ανέφερε ο Επίτροπος, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συλλέξει τα πρώτα αποτελέσματα του πιλωτικού προγράμματος για έξι χώρες και θα συντάξει τη σχετική πολιτική. Πραγματικά είναι σημαντικό ότι μη κρατικοί φορεί και οργανώσει των κοινωνία των πολιτών, όπω οι εθνικέ ε, εταιρείε και οργανισμοί, να μπορούν να υποστηρίξουν ε, την όλη διαδικασία μέσω συστάσεων και αυτό το έγγραφο είναι μια μετριοπαθή προσπάθεια γι' αυτό. Αλλά συμμετέχοντα σε τοπικό επίπεδο σε εργαστήρια και διαβουλεύσει, που από ό,τι γνωρίζουμε αυτό μέχρι τώρα δεν έχει λάβει χώρα. Δεν γνωρίζουμε σε καμία από τι έξι πιλωτικέ χώρε ότι οι εθνικοί φορεί του Εθνικού του Ερυθρού Σταυρού ή της Ερυθράς ε, ή Μισελίνου έχουν κληθεί να συμμετάσχουν στις διαβουλεύσεις. Όπως αναφέρθηκε, τώρα τρία χρόνια πέρασαν από την πρώτη σύνοδο κορυφής για τα ανθρωπιστικά θέματα, όπου ενίσχυση του συσχετισμού έχει τονιστεί από τους εμπλεκομένους φορείς και θεωρείται ύψιστη προτεραιότητα της Συνόδου Κορυφής και οι συζητήσει γύρω από τη δέσμευση να παρασχεθεί περισσότερη υποστήριξη και μέσα χρηματοδότηση στου ντόπιου φορεί ανταπόκρισης. Η συζήτηση για την ντόπια αντιμετώπιση εστιάστηκε ε, επί αυτή τη του τουλάχιστον 25% τη χρηματοδοτήσεω να δείτε σε τοπικούς και εθνικού φορείς ανταπόκρισης. ετοιμάζοντα την παρέμβασή μου ρώτησα του συναδέλφου ε, στο Διεθνή Ιθρο διότι η ελβετική κυβέρνηση και ο Ερυθρός ε, Σταυρός κινούνται σε αυτήν την κατεύθυνση. Είπαν δεν ξέρουμε ακριβώς. Μεταξύ 0,2 και 2% μιλάμε. Το να μιλάμε για 25% πόρο απέχει από αυτά τα ποσοστά. Ε, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ενδιαφέρον ότι στην στην αποστολή στον Πογκλαντές και στο Ιράκ που είναι πολυτομιακή, πολυσχηδής, οι περισσότεροι φορείς, οι τοπικοί, είπαν ότι θα καλωσόριζαν μία συνεργασία που ξεπερνά πέρα το θέμα της χρηματοδοτήσεως και πόσο κερδίζουμε από την ε, προσπάθεια που καταβάλλεται επί τόπου, μιλώντας για συνεργασία που εδράζεται επί αμοιβαίου σεβασμού δηλώσεων σαφών και σαφών συμφωνιών περί του δέον γενέστε και για ποιους λόγους γίνεται αυτό που πρέπει να γίνει. Οι τοπικοί φορείς παρέχουν υπηρεσία καθημερινά στην κοινότητά τους βάσει των αναγκών. Πραγματικά είναι η πρώτη γραμμή που ανταποκρίνεται στις καταστροφές, στις συγκρούσεις, στις σειράξεις και είναι η πρώτη γραμμή για τη δημιουργία αντοχής ε, σε επαφή με τις τοπικές αρχές. Εφαρμόζουν την ανθρωπιστική βοήθεια και την αντοξιακή βοήθεια και τη διασύνδεση αυτή μεταξύ των δύο την εφαρμόζουν επί τόπου. Ευχαριστώ όλου τους παρεμβαίνοντες. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πέντε λεπτά, τρία, πέντε λεπτά αν θέλει να, να κάνει κάποιος κάποια παρέμβαση. Η Λίντα. Ο Ζαν Λουί, θες και εσύ να πεις κάτι μετά. Πρώτα η Λίντα και μετά εσύ. Ευχαριστώ. Uh, ευχαριστώ, Ενρίκε. Ευχαριστώ τους ε, ομιλητές. Δεν είμαστε τόσοι βουλευτές um, παρόντες. Έχουμε μπει σε τρόπο λειτουργίας προεκλογικής. Αυτό δείχνει. Δεν δείχνει αδιαφορία τα ανθρωπιστικά θέματα. Τα συζητήσαμε επί σειρά ετών στην Επιτροπή μας τα ανθρωπιστικά ζητήματα ε, για τους, ε, για τους χωρίς σύνορα. Με ενδιαφέρε αυτό που άκουσα ε, ανησυχητικά αυτά που είπατε για το προσωπικό. Το θέμα της ποινικοποίηση της βοήθειας προς ανθρώπους τι γίνεται και η προστασία των εργαζομένων στον ανθρωπιστικό τομέα μας ανησυχεί. Αυτό που συνέβη στο Κοντούς δεν έγινε ε, σωστή έρευνα αυτού που συνέβη. Πρέπει αυτά να καλυφθούν αυτά τα θέματα. δύσκολη κατάσταση όταν υπάρχουν συγκρούσεις. Αν είναι σαφώς καθορισμένη ζώνη πολέμου μια περιοχή, γνωρίζει η ανθρωπιστική οργάνωση ότι άλλαξε το καθεστώς και μπορεί να αποσυρθεί. Μαζί με τους ασθενείς μπορεί να απομακρυνθεί. Αυτό έχει γίνει σε πολλές συγκρούσεις, σε πολλές σειράξεις. Εάν θεωρείται ότι ένα νοσοκομείο στεγάζει κάποιου υπόπτου, ε, θα πρέπει να μπορούν να κάνουν και οι γιατροί κάτι για του υπόλοιπου. Το θέμα των συνεχιζομένων σειράξεων. Ήρθε και Ενρίκε. Με τις ανθρωπιστικέ ε, ΜΚΟ είχαμε συναντηθεί πριν από κάποιου μήνε. Μα είπαν ότι πρέπει να διαχωρίζουμε την πολιτική από την ανθρωπιστική βοήθεια. Εμεί αυτό πιστεύουμε. Αυτοί μα είπαν το αντίθετο. Έχουμε τι λησμονισμένες κρίσει σε όλο τον κόσμο. Χρειάζονται πολιτικές λύσεις αυτέ οι λησμονημένες κρίσει. Δεν να απειλήσουμε την ανθρωπιστική κρίση επιτόπου, διότι οι πολιτικοί λησμονούν τη ρίζα του προβλήματο. Μήπω πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο να βρούμε πολιτικέ λύσει στι συνεχιζόμενες κρίσει, να δώσουμε προτεραιότητα. Ήμουνα στη Βόρεια Ουγγάντα, Φερρυπίν. Οι Νότιο Σουδανοί στον... ε, ξέφευγαν, επέναγαν τα σύνορα και ερχόταν. Δεν υπάρχει πολιτική βούληση εξέβρεση λύση. Πηδάμε από κρίση σε κρίση. Εστιαζόμαστε μια κρίση για λίγο, προχωράμε και αφήνουμε τι κρίσει να σιγοκαίνε. Και δαπανάμε χρήματα για τσίχλε κυριολεκτικά για να καλύψουμε τα κενά που έχουμε αφήσει. Πώ μπορούμε να κουβεντιάσουμε την πολιτική να συζητάμε ανθρωπιστική βοήθεια χωρίς να δούμε πολιτική απόχρωση στην ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτό είναι ένα θέμα προς προβληματισμό όλων αναφέρθηκαν η αναπάντα είχε συνέπειε τη ε, νομοθεσία. Η Voice μα είπε ότι η νομοθεσία για να σταματήσουμε την τρομοκρατία και προσπαθούμε να σταματήσουμε τα χρήματα να δίνουν χρήματα στου τρομοκράτε και αρνούνται να λειτουργούν κάποιε τράπεζε σε κάποιε χώρε. Πρέπει να κουβαλάνε μετρητά σε τεράστια ποσά οι ανθρωπιστικοί ε, εργαζόμενοι στο ανθρωπιστικό τομέα. Αναφερθήκατε στο Ιράκ και στο Ιράν. Και γίνονται στόχοι αυτοί που εργάζονται για ανθρωπιστική βοήθεια. Για ομάδε που ξέρουν τι κουβαλάνε με τριτά πάνω του για να του ληστέψουν. Δεν ξέρω, μπορεί να το σχολιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Voice μα ζήτησε να το εξετάσουμε. Εγώ μεγαλόφωνα σκεφτόμουν και έλεγα τα κρατη μέλη έχουν πρεσβείε σε δύσκολε χώρε. Θα πρέπει να στέλνουν κάποιου πόρου σε αυτέ τι χώρε. σω τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να βοηθήσουν να φτάσουν χρήματα σε ΜΚΟ που λειτουργούν νόμιμα επιτόπου σε δύσκολες κρίσεις, χωρίς να πρέπει να κουβαλάνε μαζί τους οι εργαζόμενοι ε, μετρητά. Και κάτι άλλο που είπα και στη Voice. Πάντα υπάρχει ο κίνδυνος κόπωσης των δωρητών με τόσες κρίσεις. Οι πολιτικοί να λένε τα ξέρουμε τα προβλήματα. Δίνουμε χρήματα και τίποτα δεν αλλάζει. Ένα θέμα που βρήκα ότι υπάρχει με την ανθρωπιστική βοήθεια είναι το πρόβλημα το γλωσσικό. Μιλήσαμε για τη διασύνδεση ανθρωπιστικής αναπτυξικής βοήθειας. Αν θέλετε οι πολιτικοί να ακούνε, πρέπει να μιλάει κανεί απλά. Βάζω ολόκληρο έγγραφο και σε ξεπερνάει το έγγραφο ή δεν πιάνει το νόημα. Κάθε ειδικότητα το κάνει αυτό. Η κάθε μία μιλάει δική της διάλεκτο. Ξύλινη γλώσσα, ορολογία, δυσνόητη για τον έξω κόσμο. Όταν ζητάς από το Κοινοβούλιο να εγκρίνει προπολογισμό. Όταν πολεμάς για πόρους και κινείς εναντί άλλων θεμάτων. Πρέπει οι πολιτικοί να καταλαβαίνουν ακριβώς τι εννοείς. Τι σημαίνει τον νέξους αυτή η λέξη στον απλό άνθρωπο. Αν το εξηγείς είναι απλό. Οι γυναίκες στη Βόρεια Ογκάντα είναι εκεί μακρόν. Και δεν αρκεί να του δίνουμε μακροπρόθεσμα βοήθεια. Πρέπει να υπάρχουν σχολεία για τα παιδιά, ιατρικέ υπηρεσίε μακροπρόθεσμε. Ανθρώπινη γλώσσα να βρούμε, να εξηγούμε τι γίνεται. Να αρπάζουν, να πιάνουν τα νοήματα οι πολιτικοί όταν αποφασίζουν. Και να πηγαίνει κανείς επί τόπου. Όταν δει κάποιο κάτι με τα ματάκια του δεν το ξεχνάει. Και έχω δει πολιτικού που πάνε σε επισκέψει και ανοίγουν τα μάτια του και πιάνουν το τι ακριβώ συμβαίνει. Τότε ίσω κατανοούν καλύτερα. Θα ήθελα να ευχαριστήσετε τους εργαζόμενους για σας. Τους είδαμε επί τόπου. Σε φρικτές συνθήκες πολλές φορές εργάζονται, σε δυσχερέστατες περιστάσεις. Επέλεξαν να είναι εκεί και αφήνουν τη δουλειά τους που κάνουν αλλού αφήνουν τη ζωή τους στην ομαλή και ζουν μια πολύ δύσκολη ζωή για να ανακουφίσουν ανθρώπους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη δουλειά που κάνουν οι οργανισμοί σας, οι φορείς σας. Σε ευχαριστώ Μελίντα. Θα ήθελα να ζητήσω από τον Σολουή να λάβει το λόγο όχι μόνο γιατί είναι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά διότι ο ίδιος προσωπικά Πολλές φορές παρέστη στις συνεδριάσεις μας για να μας ενημερώσει για τις διάφορες κρίσεις, καταστροφές ανά τον κόσμο. Ήταν πάντα η πρώτη φωνή που εκπροσωπούσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις νέες κρίσεις που συνέβαιναν ανά τον κόσμο. Και νομίζω ότι αξίζει να του δώσουμε τώρα το λόγο Τώρα που είναι η τελευταία συνεδρίαση πρακτικά της Επιτροπής μας και για τα ανθρωπιστικά θέματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Μακάουαν που συγκάλεσε ε, τη συνεδρίαση σε πολύ επίκαιρη στιγμή. Εγώ θα έλεγα ότι μέχρι τώρα όλα υπόθηκαν. Τα είπε και ο Επίτροπος. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, όχι μόνο για μας, αλλά για όλο το προσωπικό της ΕΚΟ, που έτυχε τη υποστήριξή σας και θέλει να σας δώσει όσο πιο δυνατόν περισσότερες πληροφορίες. Γιατί είναι επίκαιρη αυτή η συνεδρίαση. Ακούγεται σαν κάτι από αποχαιρετιστήριο, αλλά είναι μια αρχή. Διότι φέτος, όπως είπατε, ε, ε, σύντομα θα υπάρξουν ακροάσεις. Θα διοριστεί η Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διορισμός νέου επιτρόπου και η συζήτηση όπως η σημερινή θα πρέπει να μας βοηθήσει να ανοίξουμε το δρόμο για νέα ατζέντα, νέο θεματολόγιο, γιατί πολλά από τα εμπόδια, τα προβλήματα που εφήγησαν σήμερα το απόγευμα είναι γνωστά. Τα αντιμετωπίζαμε επί πενταετία. Δεν μπορούμε αένα να παραπονιόμαστε για την κατάσταση χωρίς να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Όπως ίσχυσε και με το σημερινό Κοινοβούλιο. Χρειαζόμαστε υποστήριξη του επόμενου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Χρειαζόμαστε την υποστήριξη του Κοινοβουλίου και να μας προκαλέσει το επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να μας πει τι κάνουμε, τι δεν κάνουμε, να διορθωθούμε. Να αναφερθώ σε πέντε ζητήματα τα οποία θίγησαν το απόγευμα. Επίση, η έλλειψη σεβασμού για το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό. Επικρατούσε απελπισία για μια περίοδο. Τι να κάνουμε και γινόταν παραβίασεις και έγινε ένα εργαλείο πολέμου αυτή η ε, άγνοια του Ερυθρού Σταυρού. Έγινε διεθνές ε, εργαλείο. Τελικά όλοι βαρέθηκαν. Είπαν αρκετά. Κάποια κάτι μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, μόνιμα και μη μόνιμα, ε, ετοιμάζονται να αλλάξουν. Γερμανία, Βέλγιο και Γαλλία ετοιμάζουν προτάσεις και αυτό δημιουργεί ελπίδες για πολιτική δράση, για αυξημένη προστασία του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού των ανθρωπιστικών ε, εκστρατιών που γίνονται. Υπάρχει μεγαλύτερη προστασία. Μην υποτιμάμε τον αντίκτυπο της ποινικοποίησης της ανθρωπιστικής βοήθειας. και τα αντιτρομοκρατικά μέτρα τι αντίκτυπο έχουν σήμερα στην ανθρωπιστική βοήθεια. Πιστεύουμε ότι χρειάζεται διάλογος μεταξύ της κοινωνίας των, της ασφάλειας και της ανθρωπιστικής ε, κοινότητας χρειάζεται τώρα. Δεν συνομιλούν οι δύο τομείς, δεν κατανοούν ο ένας τομέα τον άλλον. Τι έχει σημασία, να έρθουν σε επαφή ταχύτερο δυνατόν. Καταπολέμηση τρομοκρατίας είναι κάτι πολύ ουσιαστικό και κάτι πρέπει να γίνει. Ναι, δεν θα ήθελα να πω από την άλλη πλευρά, αλλά από την άλλη πλευρά αυτή είναι που είναι επιφορτισμένοι με την καταπολέμηση τη τρομοκρατία μπορεί να καταλάβουν ποια είναι η έννοια τη ανθρωπιστική δράση και τη βοήθεια, αν του το εξηγήσουμε. Το κάναμε ετοιμάζοντα την οδηγία καταπολέμηση τρομοκρατία. Υπάρχει κοινό τόπο και λύσει. Το πρώτο ήταν αυτό. Δεύτερον, τοπική αντιμετώπιση. Δεν έχουμε υψηλό, υψηλή απόδοση. Όταν συζητούμε την τόπια αντιμετώπιση, είναι πιο σημαντικό από ό,τι νομίζουμε οι τοπικοί φορείς να συμμετάσχουν, να δημιουργηθεί δυναμικό επιτόπου. να μην έχουμε μια δασκαλίστικη προσέγγιση όσον αφορά τη χωρίς ανθρωπιστικής ε, βοήθειας. Χρειάζεστε, σας δίνουμε. Ξέρουμε, δεν ξέρετε. Θα σας κάνουμε καλό, ακόμα και αν δεν θέλετε. Και άλλες δεσμεύσεις στη Μεγάλη Συμφωνία πρέπει να εφαρμοστούν. Οι δικαιούχοι να συμμετάσχουν στην ανθρωπιστική βοήθεια. Λοιπόν, πριν γίνουν επιχειρήσεις επιστροφής, Εκείνοι που έχουν χτοπιστεί δεν πρέπει να ρωτηθούν. Θέλουν να επιστρέψουν ή όχι. Πού θέλουν να επιστρέψουν, υπό ποιε συνθήκε. Πώ θα του βοηθήσουμε να επιστρέψουν. Η τοπική διάσταση είναι παρούσα. Αλλά είναι πολυσχηδή διάσταση. Αλλά ξεπερνάει τα όρια τόνωση οικονομική των τοπικών φορέων. Για την τριπλή διασύνδεση, τον τριπλό αυτό κόμβο αυτό που είπατε κυρία Μακάου, είναι πολύ σημαντικό. Μη θεωρούμε ότι δεν πρέπει να εξετάζουν την πολιτική χρειά των θεμάτων. Φαρμογή εφαρμογή παρέμβαση ανθρωπιστική στη Συρία, στην Ιεμένη, στο Ιράκ, στη Βενεζουέλα και γειτονικέ χώρε, Μπαγκλαντέ, όλα αυτά είναι ανθρωπογενείς κρίσεις. Δεν είναι φυσικέ καταστροφές. Πρέπει να έρθουμε σε επαφή με αυτού που είναι στη ρίζα του κακού. Χρειάζεται ολιστική αντιμετώπιση. Δεν αφορά χειραγώγηση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Η ανθρωπιστική βοήθεια θα συμβάλλει σε αυτή την προσέγγιση την ολιστική, χωρίς να χειραγωγείται. Έχουμε συνεννόηση με την υπηρεσία ανθρωπιστικής, εξωτερι, ε, την υπηρεσία εξωτερικής δράσης στο πώς πρέπει να χορηγείται ανθρωπιστική βοήθεια. Χρειάζεται σφαιρική προσέγγιση, πολυσχηδής προσέγγιση, συμπεριλαμβανομένης διπλωματίας, συμπεριλαμβανομένου διαλόγου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής πτυχής. Τέλος, ψηφιοποίηση και τα σχετικά προβλήματα. Συμφωνώ μαζί σου, Βόλτερ είναι μεγαλύτερη εικόνα. Μιλάμε και για καινοτομία, για χρήση νέας τεχνολογίας και όλα αυτά στην προσπάθεια καλύτερης απόδοσης στην προσπάθεια που καταβάλουμε για ανθρωπιστική βοήθεια. Να θέσουμε τάξη στους όρους και στην προσέγγιση. Χρειάζεται χρηματοδότηση. Πρέπει να δραστηριοποιηθούμε, να βρούμε νέους οικονομικούς πόρους. Συμφωνώ. Να αντιμετωπίσουμε το όλο θέμα με την εμπλοκή ίσως του ιδιωτικού τομέα. Κοιτάξτε, ευχαριστούμε πάρα πολύ από πλευράς των υπηρεσιών της ΕΚΟ. Πολλά από αυτά που υπόθηκαν θα τα διαβιβάσουμε και θα τα υπόψη στην προετοιμασία του θεματολογίου που θα υποβάλουμε στον ε, αρμόδιο επίτροπο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την πάρα πολύ εμπεριστατωμένη παρέμβαση. Θα ήθελα να δώσω το λόγο σε όποιον θέλει από τους παρεμβαίνοντες στην έδρα να λάβει το λόγο. Για δύο λεπτά όμως παρακαλώ κανατανότατο όριο ε, για να μην ξεπεράσουμε πάρα πολύ τον καιρό που είμαστε. Δύο λεπτά είμαι. Πολύ απλά θα μιλήσω. localization. Τίποτα δεν σημαίνει αυτό για μας. Συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο Υγείας και με το τοπικό προσωπικό σε κάθε χώρα. Επίσης πρέπει να δουλέψουμε με τις ε, διεθνείς οργάνωσες όπως ο Ερυθρός Σταυρός. Τον Nexus. Ένα παράδειγμα. Η ανάπτυξη του νέξου στα πλαίσια της ανθρωπιστικής βοήθειας. Στην Δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής συνεργαζόμαστε με εδώ και 10 χρόνια εδώ και χρόνια με τις δημόσιες, ε, τα δημόσια νοσοκομεία και ξέρουμε ότι είμαστε στην, ε, σε θέματα υγείας στη χώρα αυτή ο πιο σημαντικός δωρητής. Δεν υπάρχει κανένας να συνεχίσει το έργο μας ή να κάνει αυτό που κάνουμε εμείς. Και πρέπει να πω ότι τα στάνταρ είναι τα ελάχιστα δυνατά. Αλλά δεν υπάρχουν ε, κοινοτικά κονδύλια, κυρίως στον τομέα της υγείας και μέσα συμπληρωματικά και εκφράζουμε την ανησυχία μας για την κατάσταση αυτή δεν υπάρχουν ούτε εθνικά ούτε διεθνή κονδύλια διαθέσιμα. Τώρα, στι επιθέσει προ νοσοκομεία. Ξέρω ότι υπάρχουν κάποιε πρωτοβουλίε, αλλά πρέπει να πω και πάλι ότι επιτόπου δεν υπάρχει αξιοπιστία όταν συμβεί κάτι τέτοιο και δεν υπάρχει και λογοδοσία. Πολλές φορές γίνονται ε, και υπάρχουν και κατηγορίες εναντίον μας ότι δεν σεβόμαστε κάποιους κανόνες. Αυτό λοιπόν το αναφέρω διότι δεν έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Και κάτι άλλο. Αυτό που είναι σημαντικό σε αυτές τις επιθέσεις δεν είναι ότι εμείς είμαστε εκεί και μπορούμε να κινδυνεύσουμε. Το σημαντικό είναι ότι τα άτομα δεν έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας μετά από αυτά που συμβαίνουν. Σας ευχαριστώ για την ε, ανθρωπιστική διάσταση και τη διάσταση της ασφάλειας. Σημειώσαμε αυτά που είπατε. Γεγονός είναι όμως ότι κάθε στρατηγική που θα εφαρμόζεται θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τις δυναμικές που υπάρχουν και που επικρατούν ε, επιτόπου. Γιατί μια τέτοια στρατηγική προλαμβάνει τον εξτρεμισμό και την τρομοκρατία. Και είναι σημαντικό γιατί πρέπει, αυτό θα επηρεάσει και τις προτεραιότητες για την τοπική διάσταση, το localization. Ε, κυρία Μακάβαν, σημειώνω αυτό που είπατε ε, για τη γλώσσα που χρησιμοποιούμε και το ότι θα πρέπει να μπορώ να εξηγήσω αυτά που κάνω και στη γιαγιά μου. Όμως ε, για την τοπική διάσταση πρέπει να σας πω το εξής. Πολλές φορές στις ανθρωπιστικές κρίσεις που αντιμετωπίζουμε και στις οποίες ε, παρεμβαίνουμε δεν υπάρχει κεντρική κυβέρνηση, υπάρχουν μόνο τοπικές κοινωνίες. Οπότε με αυτόν τον όρο αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι θέλουμε να βοηθήσουμε τις τοπικές κοινωνίες μακροπρόθεσμα να ε, αναπτύξουν τις ικανότητες τους ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις ε, προκλήσεις που, που αντιμετωπίζουν. Θεωρούμε λοιπόν ότι όλο και περισσότερα ε, κράτη-μέλη βλέπουμε μάλλον ότι πιστεύουν ότι μπορούν ε, ε, να μην λογοδοτήσουν ποτέ για πράξεις τους, για προβλήματα που τα ίδια έχουν προκαλέσει. Η λύση λοιπόν σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να προέλθει από, τους, από τις ανθρωπιστικές οργανώσεις. Πολλές φορές ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια τέτοια προσδοκία επαναλαμβάνω και από αυτό το βήμα ότι δεν μπορεί κανείς να περιμένει οι ανθρωπιστικές οργανώσεις να λύσουν όλα τα προβλήματα. Συμφωνώ απόλυτα ότι σε μια πρώτη φάση μπορεί η ανθρωπιστική βοήθεια να δίνεται με έναν δασκαλίστικο τρόπο, με έναν πατερναλιστικό τρόπο. Όμως αυτό που πρέπει να ε, σημειώσουμε είναι ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει Αφενό να αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια, ταυτόχρονα όμω να συνοδεύεται και από πιο αυστηρού κανόνες. Δεν ε, έχουμε αρκετό χρόνο, αλλά ε, υπάρχει για παράδειγμα ο Δανέζικος ε, Ερυθρός Σταυρός, ο οποίος έχει έλθει σε συμφωνία με, με μία από τις τέσσερις μεγάλες λογιστικές ελεγκτικές εταιρείες, κάτι που τον έχει βοηθήσει για την καλύτερη διαχείριση των οικονομικών του. Ευχαριστώ πολύ. Να πω κάτι για αυτό που είπε η κυρία Μακάβαν για την πολιτική δράση. Εμείς θέλουμε οι πολιτικοί να λύσουν τις πολιτικές κρίσεις. Αυτό που λέμε όμως ταυτόχρονα είναι ότι δεν θα πρέπει οι πολιτικοί να παρέχουν την ανθρωπιστική βοήθεια. Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις θα πρέπει να αναλάβουν την ανθρωπιστική βοήθεια για ανθρωπιστικούς σκοπούς και οι πολιτικοί ε, άνδρες και γυναίκες θα πρέπει να επιληφθούν των πολιτικών κρίσεων. Προφανώς εμείς ως ανθρωπιστικές οργανώσεις δεν μπορούμε να δώσουμε πολιτικές λύσεις. Γι' αυτό και καλούμε τους πολιτικούς να κάνουν τις απαραίτητες κινήσεις. Θέλω να πω ότι σε τελική ανάλυση στην ε, παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας θα γινόμαστε πιο αποδεκτοί από τους, από τους αποδέκτες της ε, βοήθειάς μας αν μας αντιλαμβάνονται πραγματικά ως ανθρωπιστικές οργανώσεις. Δεν έχουμε καμία δουλειά εμείς οι ανθρωπιστικές οργανώσεις ούτε να συλλέγουμε μυστικές πληροφορίες, ούτε να κάνουμε πολιτικές παρεμβάσεις, ούτε τίποτα τέτοιο. Εμείς, τη δουλειά μας, ανθρωπιστική βοήθεια. Και για να γίνει αυτό χρειάζεται διάλογος. Ακόμη και αν η μία ή η άλλη πλευρά χαρακτηρίζεται ως τρομοκρατική. Είναι σημαντικό να ενισχύσουμε και το διάλογο μεταξύ μας για την ανθρωπιστική ενώ βοήθεια σε σχέση με την ε, αντιμετώπιση τρομοκρατικών απειλών. Πρέπει να ενισχυθεί ε, ο διάλογος. Εμείς θα προσκαλούσαμε, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι, την Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, εξετάσει τη δυνατότητα να δοθούν εξαιρέσεις ανθρωπιστικές σε εκείνους που έχουν αποδείξει στην πράξη ότι ακολουθούν και πληρούν όλα τα κριτήρια. Τέλος. Που θεωρώ ότι είναι και πάρα πολύ σημαντικό. Μιλάμε για πληθυσμούς και τη δική μας λογοδοσία απέναντι σε αυτούς μπορώ να σας πω ότι έχουμε εκδώσει εσωτερικά κατευθυντήριες γραμμές ακριβώς για αυτή τη λογοδοσία απέναντι στους πληθυσμούς που βοηθάμε. Τώρα θα πρέπει και εγώ να παρουσιάσω τα συμπεράσματα αυτής της ε, συζήτησης που είναι στα πλαίσια της ακρόασης για την ανθρωπιστική βοήθεια και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Δεν θα μιλήσω για 45 λεπτά, ούτε καν 5. Δύο λεπτά μόνο. Πρώτα απ' όλα διότι πιστεύω ότι σήμερα που ευχαριστούμε ως μόνιμος εισηγητής για το θέμα αυτό θα πρέπει να ευχαριστήσω όλους όσους με βοήθησαν στα πλαίσια της Επιτροπής Ανάπτυξης. Να ευχαριστήσω και τον Μανουέλ και την Τζοάνα και τις διάφορες πολιτικές ομάδες που πολλές φορές έλαβαν το λόγο για να εστιαστούμε στις διάφορες ανθρωπιστικές κρίσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Βρίσκαμε σε στιγμή αλλαγή. θα γίνουν ευρωεκλογέ σε δύο μήνες, σε τρεις μήνες, συγγνώμη, πιστεύω ότι στις διάφορες παρεμβάσεις τονίστηκε η ανάγκη στο επόμενο κοινοβούλιο, στους επόμενους συναδέλφους, να πούμε ότι ανησυχούμε διότι υπάρχουν σε σχέση με τις ε, αρχές ε, που πρέπει να διέπουν την ανθρωπιστική βοήθεια και τη διεθνή νομοθεσία διάφορες ε, παραβιάσεις και ερωτηματικά. Θα πρέπει λοιπόν να λάβει δεσμεύσεις το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να διαθέσει τα κατάλληλα μέσα ώστε σε ένα κόσμο που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ανθρωπιστικής κρίσης να κάνει κάτι για να διορθώσει την κατάσταση και να χρησιμοποιήσει με πιο αποτελεσματικό τρόπο τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Αλλά θα πρέπει να ανοίξουμε τα μάτια μας και να δούμε με μεγάλη καθαρότητα τα φαινόμενα τα οποία επαναλαμβάνονται και δεν υπήρχαν στην ε, σημερινή τους διάσταση, όπως παραδείγματο χάρη την παρέμβαση των ε, γιατρών χωρίς σύνορα. Σε μια συνάντηση που είχαμε με τους γιατρούς του κόσμου σήμερα, είδαμε ότι στις κρίσεις, στις μακροπρόθεσμες, αυτής της ε, ανθρωπιστικής κρίσης αυξάνονται οι ψυχικές ασθένειες με μεγά... σε μεγάλο βαθμό. Θα πρέπει λοιπόν να καταβληθούν προσπάθειες στα διάφορα συστήματα υγείας για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή την κατάσταση όλοι μαζί διότι ο τρόμος, ο φόβος, η καταστροφή, η ανάγκη να διαφύγει κάποιος μπορεί να δημιουργήσει τρομερά ψυχικά προβλήματα. Νομίζω ότι έχει γίνει συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα και θα πρέπει να συνεχιστεί για τον σχέση μεταξύ της παροχής της ανθρωπιστικής βοήθειας σεβόμενη την διεθνή νομοθεσία, την συνένεση και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά όντας συγχρόνως ενεργεί ώστε να μπορούμε να προβλέπουμε διενέξεις, σειράξεις, συγκρούσεις και να κάνουμε ένα βήμα πριν να χειροτερέσει κατάσταση. Θα πρέπει να βρούμε ένα σημείο ισορροπίας. Δεν μπορούμε πάντα να έχουμε το 50 50 θα πρέπει να σεβόμαστε τις ιδιαιτερότητες της ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά δεν θα πρέπει να είμαστε κοντόφθαλμοι. Δηλαδή, να αναγνωρίσουμε ότι προβλήματα που δεν μπορούμε να τα λύσουμε μέσω της ανθρωπιστικής βοήθειας, να χρειαστεί να τα λύσουμε με πολιτική βοήθεια. Τι σημαίνει ότι το επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να προωθήσει μια πιο ενωμένη πολιτική Ευρώπη και όχι να οδηγήσει σε διαχωρισμούς. Τώρα, το απόγευμα είναι υπέροχο σήμερα. Σαν να είμαστε στην Κρήτη, στη Μαδρίτη και όχι στις Βρυξέλλες με τον καιρό που κάνει. Δεν θα διαρκέσει όμως αυτός ο καλός καιρός. Κακά νέα έχω να σας πω. Την επόμενη εβδομάδα έρχονται κάποιοι δικοί μου προσκεκλημένοι και από ό,τι είδα στις Βρυξέλλες έχουμε 10 μέρες βροχή από αύριο. Λοιπόν, εάν έχετε την δυνατότητα να πάτε να επωφεληθείτε από τον καλό καιρό στην πλατεία του Λουξεμβούργου. Βεβαίως αφού ακούσουμε πρώτα τι έχουν να μας πούν οι συνάδελφοι που πήγανε στην αντιπροσωπεία στην Γκάμπια. Θέλουμε να υποφεληθεί όλο ο κόσμο από την ανθρωπική βοήθεια, αλλά δεν μα είπε κανεί να μην υποφεληθούμε κι εμεί από τον καλό καιρό σήμερα το απόγευμα. Α το προσπαθήσουμε λοιπόν. Α ακούσουμε όμω πρώτα του συναδέλφου που πήγαν στην επίσκεψη αυτή στην Κάμπια. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Okay, colleagues. Enrique. Ορίκε, μίλησε για τον υπέροχο καιρό. Α τελειώσουμε γρήγορα τη συνεδρίαση. Σημείο 14 ανεβλήθη. Το ανακοίνωσα άλλωστε. Τελευταίο σημείο είναι το 15. Ενημέρωση της αποστολής της Επιτροπής Ανάπτυξης εις Γκάμπιαν. Ο Νόρμπερτ Νόιζερ έχει το λόγο που ηγήθηκε στην αντιπροσωπεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Λίντα. Νομίζω ότι ήταν επιτυχέστατη η αποστολή. Είδαμε μεγάλη πρόοδο. Πολλές επιτυχίες. Η αντιπροσωπεία της Επιτροπής Ανάπτυξης στην Κάμπια έγινε πέρσι το Δεκέμβριο. Γιατί πήγαμε. Θέλαμε να δούμε τη μετάβαση της χώρας προς τη δημοκρατία. Μετά την ήττα του Προέδρου Τζαμέ που προκάλεσε έκπληξη το Δεκέμβριο του 2016 στις προεδρικές εκλογές. Μετά από 22 χρόνια δικτατορία ιτήθηκε. Η άνοδος του Αντάμα Μπορώ στην εξουσία τον Ιανουάριο 2017 του Προέδρου της Αντιπολιτεύσεως και οι δημοκρατικές εκλογές και κοινοβουλευτικές τον Απρίλιο οδήγησαν σε αύξηση της αναπτυξιακής βοήθειας στη μικρότερη χώρα της ε, Αφρικανικής Υπήρου και μία από τις λιγότερο ανεπτυγμένες στον κόσμο. Είναι στην 173η θέση από τις 188 χώρες η Γκάμπια όσον αφορά την ε, ανάπτυξη, την ανθρώπινη ανάπτυξη. 63,5% πάνω από το μισό του πληθυσμού στην Γκάμπια είναι σε ηλικία μικρότερη των 25 ετών. Η αιτήσια ανάπτυξη πληθυσμού είναι στο ρυθμό 3,2% η οικονομία ουσιαστικά είναι αγροτική οικονομία. Η Γεωργία έχει περίπου το 30% του ΑΕΠ. Η επίσκεψη εστιάστηκε επί της νεολαίας των θέσεων εργασίας και αποτελεσματικής των προγραμμάτων EDF και Trust for που σχετιζόταν με την νεολαία και απασχόληση και τη μετανάστευση και την αύξηση της δημοκρατικής διακυβέρνησης, την επίλυση μάλλον των προβλημάτων όσον αφορά την ε, δημοκρατική διακυβέρνηση της χώρας. Ήταν ε, φορτωμένο το πρόγραμμα, λίγες μέρες. Είχαμε πάρα πολλέ συναντήσεις. Συναντήσαμε πάρα πολλούς συνομιλητές, ευρύ φάσμα εκάλυπταν. Και κάναμε, επισκεφτήκαμε και διάφορα έργα και προγράμματα. <coughs> Ενημερωθήκαμε. Δεν συναντήσαμε τον πρόεδρο Μπόρο, συναντήσαμε τον αντιπρόεδρο Ντάμπο. Ο πρόεδρος δεν ήταν στην Πανγιούλ την ημέρα που πήγαμε. Συναντήσαμε και τον πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης και αρκετούς υπουργούς της κυβέρνησης. Όλες οι συναντήσεις ήταν εγκάρδιες, ανοιχτές, δημιούργησαν θετικές εντυπώσεις όσον αφορά το νέο πολιτικό τοπίο. Ο θετικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Ενώσης υπογραμμίστηκε ξεκάθαρα. Πολύ ενημερωτική συζήτηση στο κοινή Τραπέζης διεξήχθη, εστιάθηκε επί της δημοκρατικής μετάβασης, μετάβαση στο μέτς δικαιοσύνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα θέματα των φύλων, ο ακροτηριασμό ε, των γυναικών, των γενετικών οργάνων των γυναικών συζητήθηκε. Μετά πήγαμε τη δεύτερη μέρα εκτός πρωτεύουση σε διάφορα έργα. Πήγαμε και στη γέφυρα Τρανσγκάμπια, 200 χιλιόμετρα ανατολικά της Μπαντζούλ, η πρώτη γέφυρα που ε, διασχίζει, ε, διασχίζει, γεφυρώνει τον ποταμό Γκάμπια ε, και θα είναι ε, σύντομα έτοιμη για αν, άνοιξε την κυκλοφορία. Οι πρόεδροι της Γκάμπιας και της Σενεγάλης ε, εγκαινιάζουν τη γέφυρα που είναι διασυνοριακή. Η γέφυρα ε, είναι οικονομική στρατηγική σημασίας. Συνδέει τα βόρεια τμήματα της Γκάμπια και της Σενεγάλης. Η γέφυρα χρηματοδοτήθηκε από την Τράπεζα Αφρικανικής Ανάπτυξης, αλλά η οδική κατασκευή α, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετανάστευση. Μετά τη μετάβαση μειώθηκε η μετανάστευση ε, από δημία από την Γκάμπια. Όταν πήγαμε 4.000 μετανάστες επέστρεψαν. Οι περισσότεροι από τη Λιβύη και κάποιοι από κάτι μέτρη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Η βοήθεια παρέχεται για αυτούς που επιστρέφουν περίπου 4 εκατομμύρια από το καταπίστευμα της Ευρωπαϊκής Ενώσης για επανένταξη αλλά κατά διάρκεια των συζητήσεων με Γκαμπιανούς που επέστρεψαν πρόσφατα είπαν ότι χρειάζεται ε, πιο μακροπρόθεσμη υποστήριξη και βοήθεια για την επανένταξη πέρα από την εντολή που έχει δοθεί στον αρμόδια φορέα. Το πολιτικό κόμμα και η κατάσταση ε, ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα βελτιώθηκε πολύ μετά την μετάβαση, μετά την αλλαγή. Έλλειψη οικονομικών ευκαιριών είναι η μεγαλύτερη αιτία της μετανάστευσης τώρα. Κάποια σχόλια για οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις. Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει προβλήματα σε όλους τους τομείς ανάπτυξης εστιάζεται ιδιαίτερα στην υγεία, στην παιδεία, τη γεωργία. Μέσω εθνικών αναπτυξιακών σχεδίων για την περίοδο 2018-2021. Η υποστήριξη για τις γυναίκες σημειώθηκε και ενθαρρύνθηκε σε πολλές από τις σκέψεις. Και χρηματοδοτούμε προγράμματα για δικαιώματα των παιδιών, δημιουργία λεσχών μητέρων να προωθηθεί η παρακολούθηση μαθημάτων στα σχολεία και η προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών. Υποστήριξη από διεθνεί εταίρου, συμπληρωμένε τη Ευρωπαϊκή Ένωση για υποδομέ, είναι κάτι που έγινε αποδεκτό. Θεωρείται πολύ επικοδομητικό για την υποστήριξη τη ανάπτυξη. Τα μέλη επισκέφθηκαν τον τόπο κατασκευή τη γέφυρα τη Τρανσγκάμπια που μπορέσαμε να την περάσουμε πεζή, τη γέφυρα. Και αναπτυξιακή βοήθεια τη Ευρωπαϊκή Ενώση χρηματοδοτεί την κατασκευή και των διάφορων ε, δρόμων που διασυνδέουν τη χώρα με τη γέφυρα. Κάποια συμπεράσματα. Πολιτική βούληση στη χώρα είναι προφανή στη χώρα. Εργάζεται, συνεργάζεται με τους διεθνείς εταίρους πολύ καλά η κυβέρνηση για να μπορέσει να πετύχει προτεραιότητε. προτεραιότητες. Συνεχίζεται η πρόοδος, αντιμετωπίζει όμως πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα σε όλου τους αναπτυξιακούς τομεί με περιορισμένες δυνατότητες που έχει η κυβέρνηση και οι δημόσιες υπηρεσίες να μπορέσουν να πετύχουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες. Στα τελικέ συναντήσεις είδαμε ότι πέρα από την οικονομική υποστήριξη χρειάζεται πολιτική δέσμευση μεγάλη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε επίπεδο κοινοβουλευτικό για την υποστήριξη της μετάβασης, να ενθαρρυνθεί ο διάλογος και να γίνει ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με του πολιτικού τη Γκάμπια και να επισκεφθούν οι πολιτικοί της ε, και η επίσκεψη πολιτικών της Γκάμπια στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ήταν ένα επιτυχές πρώτο βήμα. Για τα αποτελέσματα. Βασικό πολιτικό αποτέλεσμα και συμπέρασμα. Και δράση πρέπει να ακολουθήσει. Θα πρέπει πραγματικά να δούμε ότι υπάρχει πολιτική βούληση στη χώρα. Πρέπει να ενθαρρυνθεί με οικονομική και μη οικονομική υποστήριξη και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργηθούν δυνατότητες στη χώρα. Η ασφάλεια εφοδιασμού σε τρόφιμα είναι ένα πρόβλημα. Βραχυπρόθεσμη υποστήριξη και μακροπρόθεσμη υποστήριξη για αναζωογόνηση του γεωργικού τομέα πρέπει να είναι ένα στόχος. Τα προγράμματα Trust for είναι θετικά. Χρειάζεται βοήθεια για οικονομική υποστήριξη για τους νέους Χρειάζεται καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση για υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων και θα πρέπει να υπάρχει σωστή εκπαίδευση στη χώρα ε, μέσω κατοίκων της Γκάμπια που έχουν εκπαιδευτεί σωστά. Αναπτυξιακά προγράμματα θα πρέπει να αξιολογηθούν για ματοπρόθεσμα αποτελέσματα και βιωσιμότητα και τα επιτυχέστερα προγράμματα να αυξηθούν σε κλίμακα για να υπάρξει πρόοδο σε μεγάλη κλίμακα στη χώρα. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εξετάσει εκ του σύνεγγυ την αξιολόγηση έργων που χρησιμοποιούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη και κατά πόσο πετυχαίνουμε του αναπτυξιακού στόχου μέσω τη χρηματοδοτήσεω. Και ελπίζουμε την επόμενη περίοδο το Κοινοβούλιο και ο λαό τη Γκάμπια ε, να κινηθούν προ αυτήν την κατεύθυνση. Ευχαριστώ, Νόρμπερτ. Άκουσα όλοι που πήγαν στην αποστολή να πούνε ότι ήταν θετικά και έχουμε θετικά αποτελέσματα. Έχουμε την υπηρεσία εξωτερική ε, δράση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι παρούσα. Λακωνικότατη, αν μπορείτε να αισθανθείτε. Τώρα με τυφλώνει και ο ήλιο. Ναι, ανεβοκατεβαίνανε και τα στόρια. Ε, σύντομα, λοιπόν. Παρακαλώ. Και πρέπει να προλάβω και το τρένο μου. Να πάω στο Λονδίνο σύντομα. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω την αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκ μέρους της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην, στην Ταμπούλ. Ε, ε, είναι, ήταν πραγματικά μια επίσκεψη που έδωσε, που έστειλε το μήνυμα ότι δεν έχουμε ξεχάσει την ε, Γκάμπια. Ξέρετε ότι από την αλλαγή της κυβέρνησης οι σχέσεις μας με τη χώρα αυτή έχουν ενισχυθεί Θέλω να αναφερθώ σε κάποια σημεία. Η Γκάμπια υπέγραψε την ε, εμπορική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικής Αφρικής. Επίσης ε, ε, υπέγραψε και την συμφωνία για την αλληλεία με τις δυτικοαφρικανικές χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει την προσήλωσή της στο, στην υποστήριξη της μεταρρυθμιστικής ατζέντα της νέας κυβέρνησης της ε, Γκάμπια και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Πρόσφατα οι ακροάσεις, ε, ξεκίνησαν οι ακροάσεις στην Επιτροπή Συμφωλίωσης. Η Γκάμπια έχει πλέον ορίσει έναν εκπρόσωπο για τα θύματα. Επίσης, πρόσφατα συστάθηκε στη χώρα Εθνική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η οποία σημείωσε σημαντική πρόταση ε, πρόοδο όταν και διορίστηκαν οι επίτροποι. Επίσης έχουμε ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση του τομέα ασφαλείας που ήταν αργή μέχρι σήμερα, αλλά πλέον φαίνεται να μπαίνει ε, με ταχύτερους ρυθμούς. Ε, ελευθερία έκφρασης, αυτό ήταν ένα από τα, μακροπρόθεσμα, από τα μακροχρόνια προβλήματα της χώρας. Ξέρετε ότι το 2018 η Γκάμπια ανέβηκε 21 θέσεις στον δίκτυο για την ελευθερία της έκφρασης. Επίσης γίνεται διαβούλευση με ε, τους... Ε, εμπλεκόμενους φορείς με, τις, ε, κοινωνία, με την κοινωνία των πολιτών για το νέο σύνταγμα της χώρας το οποίο θα μπει σε δημοψήφισμα στις αρχές του 2020. Γενικά η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, εκφράζει την ικανοποίησή της για τις θετικές εξελίξεις ε, που έχουμε σε μια ε, ευρύτερη πορεία που ε, θα μας οδηγήσει σε μια πραγματική δημοκρατική μεταρρύθμιση της χώρας. Ο κύριο Στάλμαν από την ε, Γενική Διεύθυνση. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο για να μπορέσουμε να επαφεληθούμε από τον ήλιο. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την ε, και Επιτροπή για τον Επαγγελματισμό και για την πάρα πολύ ατμόσφαιρα που επικρατούσε στα πλαίσια της αντιπροσωπείας. Νομίζω στα πλαίσια της νέας αυτής δημοκρατίας Τέτοιου είδους αποστολές αποδεικνύουν ότι από πολιτικής πλευράς είναι πάρα πολύ καλά, θετικά παρούσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως συγκεκριμένη περίπτωση. Και σε δύο χρόνια από μια αντιπροσωπεία που είχε να χειριστεί 33 ε, εκατομμύρια ευρώ, σε δύο χρόνια φτάσαμε στα 330 εκατομμύρια. Δεκαπλασιάστηκε λοιπόν το κονδύλι το οποίο διαθέσαμε για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε αυτή την ε, δημοκρατία. Τα μέλη της αποστολής λοιπόν ε, υπογράμμισε πόσο σημαντική ήταν αυτή η προσπάθεια και θα ήθελα και εγώ να τα ευχαριστήσω διότι πρέπει να πω ότι ήταν εξαιρετική η εργασία που επιτέλεσαν. Ήθελα επίσης να συμφωνήσω με το συμπέρασμα ότι ίσως ε, η, για την ανάπτυξη της χώρας αυτής αποτελεί τροχοπέδι το ότι ο δανεισμός ανέρχεται στο 130% του ΑΕΠ. Πρέπει να πω ότι γι' αυτό και εμείς στα πλαίσια της συνεργασίας μας τα δύο τελευταία χρόνια προσπαθούμε να δώσουμε οξυγόνο στα οικονομικά της χώρας αυτής και επίσης τα θέματα των ε, υποδομών, ο συντονισμό, σε θέματα υποδομών για να χτιστεί αυτή η γέφυρα, αυτή το κοινό δίκτυο και έχουμε και ενεργειακά σχέδια που αφορούν ε, για όλα τα σχολεία και όλα τα κέντρα υγείας της χώρας προβλέπουμε ηλιακούς, ηλιακά πανό, ώστε να μπορέσουν όλα τα υγειονομικά κέντρα και τα σχολεία να έχουν θέρμανση. Επίσης, θα πρέπει να δώσουν, ξαναδώσουμε εμπιστοσύνη στους νέους σε σχέση με τη δημοκρατία και να δείξουμε πώς λειτουργεί αυτή η δημοκρατία. Γι' αυτό σε θέματα απασχόλησης επικεντρωνόμαστε επίσης στα πλαίσια του πολιετούς χρηματοδοτικού πλαισίου, Continuer, euh, pour... τα δέκατα του τέτοιου πλαισίου, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης και να προσφέρουμε βιώσιμες λύσεις σε θέματα απασχόλησης, κυρίως στους νέους και στην οικονομία της χώρας αυτής. Γενικότερα ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Βλέπουμε λοιπόν πρόοδο σε αυτή τη χώρα και από οικονομική πλευρά και από ανθρωπιστική πλευρά και από πολιτική. Ευχαριστούμε, Νόρμπερτ, για αυτή την έκθεση. Φτάσαμε τώρα στο τέλο των εργασιών μας. Στα διάφορα δεν έχουμε τίποτε. Επόμενη συνεδρίαση 18 Μαρτίου στις 3 η ώρα το απόγευμα. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Έχετε ακόμη χρόνο για να επωφεληθείτε από τον ήλιο. Ξέχασα να πω ότι στις 4 Μαρτίου έχουμε μια κοινή συνεδρίαση με την ΑΦΕΤ και ψηφοφορίες. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Καλό βράδυ αυτή την ε, τελευταία μέρα του αναπάντεχου καλοκαιριού στις Βρυξέλλες.